Okay, friends, uh, we won't be that many. Αγαπητοί φίλοι, δεν είμαστε πολύ παρόντες σήμερα. Ας προσπαθήσουμε να εργαστούμε αποτελεσματικά και να ε, εξετάσουμε την ημερήσια διάταξη όπως έχει προγραμματιστεί. Η ημερήσια διάταξη μπορεί να υιοθετηθεί με τις εξής τροποποιήσεις. Δύο θέματα, το 7 και το 8 Το πρώτο για το EGF και το δεύτερο για τη ΣΥΤΑ αναβάλλονται για τις 8 Δεκεμβρίου. Δεν θα ψηφίσουμε κατά τη σημερινή συνεδρίαση. Διερμηνία διατίθεται σε όλες τις γλώσσες εκτός από εστονικά. Υπάρχει κάποια υποστήριξη ε, για κάποιους από εσά. Ε, Κροατικά και γοηδελικά επίσης δεν ε, διατίθενται. Τούτου λεχθέντος περνάμε στο σημείο 3 της ημερησίας διάταξης. Προσέγγιση των ε, κανόνων και διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά ε, τις ε, απαιτήσει ε, περί προσβασιμότητας ε, για τα προϊόντα και τι υπηρεσίε. Για να είναι προσβάσιμη και η σημερινή συζήτηση στα πρόσωπα με αναπηρία, προβλέπεται διερμηνία στην νοηματική. καθώς ε, και μετατροπή σε γραπτό κείμενο. Θα δώσω σε λίγο τον λόγο στον ε, εισηγητή. Η Επιτροπή Απασχόλησης έχει αποκλειστική ε, αρμοδιότητα για κάποιες από τις διατάξεις. Πολλές όμως διατάξεις καλύπτονται από κοινού από την Επιτροπή ΙΜΚΟ και εμάς. Το υπόλοιπο το τμήμα του παρατήματος 1 θα συζητηθεί κατά μια κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Απασχόλησης Μεταφορών και Εσωτερικής Αγοράς. ΙΜΚΟ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Άνταμ Κόσα, που θα μας εξηγήσει γιατί και πώς ε, η οδηγία αυτή μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εξαλείφοντας ε, εμπόδια, έχετε λοιπόν το λόγο κύριε Κώσα. Ευχαριστώ πολύ Κυρία Πρόεδρε, διαβάσατε τον τίτλο του σχεδίου οδηγίας, ο οποίος δείχνει σε τι βαθμό πρόκειται για τεχνικής φύσης ζήτημα. Η Επιτροπή μας ε, αντιμετωπίζει πολύ δύσκολο έργο. Ε, θα ήθελα όμως ε, να τονίσω τα βασικά θέματα. Καταρχάς, είχαμε διάφορες διαβουλεύσεις ε, έχουμε συνομιλήσει με εμπειρογνώμονες και προφανώς ε, έχουμε ασχοληθεί με κάποια από τα θέματα αυτά επανειλημμένα. Θα ήθελα λοιπόν ε, να τονίσω το εξής. Έχουμε μια νομοθετική πρόταση. Πολλοί συναδελφοί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ασχοληθεί με τα θέματα αυτά εδώ και αρκετό καιρό. Άρα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να λάβουμε υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σειρά της έχει κυρώσει το πλαίσιο αυτό. Βλέπουμε ότι πρόκειται για ζητήματα νομοθετικού χαρακτήρα που διευθετούνται μέσω κανονισμών. Άρα μπορεί ενδεχομένως να υπάρχει αντίφαση μεταξύ των διαφόρων κανονισμών. Γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να άρουμε αυτές τις αντιφάσεις. Όπως σας είπα, πρόκειται για ένα ε, χαρτοφυλάκιο τεχνικού χαρακτήρα και έχουμε λάβει 230 τροπολογίες περίπου. Το ζήτημα αυτό μπορεί να διευθετηθεί κατά ένα τρόπο μόνο, μέσω συνεργασίας και συνεννόησης. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο μέχρι τέλους. Εγώ είμαι πρόθυμος να αποσύρω τις ε, τροπολογίες μου για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Το δεύτερο ζήτημα που βλέπω είναι το εξής. Αν λάβουμε υπόψη την ομοθετική διαδικασία και τους τριμερείς διαλόγους, εξαναρχίζει ο μιλητής και ρωτά κατά πόσο υπάρχει θέμα με τη διερμηνία. Ωραία. Επαναλαμβάνω, λαμβάνοντας υπόψη τους ε, τριμερείς ε, διαλόγους, μετά το 19 θα τεθεί σε εφαρμογή αυτό το κείμενο και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποιες θα είναι οι τεχνικές αλλαγές μέχρι τότε. Άρα θα πρέπει να εγκρίνουμε έναν ευέλικτο κανονισμό, ο οποίος να αντιστοιχεί στις καινοτομίες που θα ανακύψουν μέχρι τότε. Το τρίτο ε, ζήτημα αφορά τη σχέση αυτού του κειμένου με τις υπηρεσίες στον οπτικοακουστικό τομέα, όπου αυτή τη στιγμή γίνεται ένα νομοθετικό έργο Δυστυχώς όμως δεν είναι συντονισμένες οι προσπαθίες μας. Προσπαθούμε να προσέξουμε και να βρούμε και άλλα μέσα, δηλαδή τα intergroup. Να συντονιστούμε λοιπόν, γιατί πρόκειται για δύο αλληλένδετα ζητήματα. Τώρα θα ήθελα να φτάσω σε ιδιαίτερα ζητήματα σε σχέση με το σήμα Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να μην αναχαιτήσουμε τη χρήση των καινοτόμων προϊόντων και παράλληλα να μπορούν όσοι έχουν κάποια αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα καινοτόμα προϊόντα. Επίσης, δεν θα πρέπει να υπάρχει αποκλεισμός ανθρώπων από την κοινωνία. Εάν εγκρίνουμε έναν πολύ συσταλτικό κανονισμό, αναρωτιέμαι κατά πόσο αυτό δεν θα είχε αντίκτυπο στην καινοτομία. Νομίζω ότι μία πολύ συσταλτική λύση θα θέσει σε κίνδυνο την καινοτομία. Γι' αυτό θα πρέπει να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο ζητήματα, ε, δηλαδή την καινοτομία και την ε, προσβασιμότητα των αμαία. Θα πρέπει κάθε προϊόν να είναι προσβάσιμο για όλες τις ομάδες της κοινωνίας. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε το ζήτημα και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση αντιμετωπίζω ορισμένα προβλήματα με το ενιολογικό πλαίσιο του κειμένου έστειλα και τροπολογίες σε σχέση με τους ορισμούς. Θα πρέπει να γίνει μία διάκριση μεταξύ βιομηχανικών χρήσεων και χρήσεων αποστεριόρι γιατί είναι διαφορετική η ευθύνη. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για ευθύνη του παραγωγού, ενώ στην άλλη περίπτωση αφορά τους φορείς. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτές τις πολλαπλές ευθύνες. Θα πρέπει επίσης να ορίσουμε και τις, ε, τις ε, λειτουργικές αποδόσεις, τη λειτουργική απόδοση δηλαδή τα προϊόντα θα πρέπει να δούμε μέχρι πού θα είναι προσβάσιμα, αλλά δεν θα ορίσουμε τον τρόπο προσβασιμότητας, γιατί οι τροπολογίες που θα υποβάλουμε ήδη θα είναι ξεπερασμένες σε δύο χρόνια με βάση τις νέες δυνατότητες που διαγράφονται. Επίσης, θα πρέπει να εξευρεθεί μία λύση σε σχέση με την εξέταση των προϊόντων και των υπηρεσιών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την δυναμική και τις δυνατότητες των νέων προϊόντων. Θα επεξεργαστώ και άλλες τροπολογίες. Θα πρέπει οι κανόνες που διέπουν τα προϊόντα, τα αγαθά και τις υπηρεσίες να μην αποτελέσουν φόρτο για τους παραγωγούς. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει και η συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρίες στο νομοθετικό έργο. Επίσης, κάθε προϊόν θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από όλες τις ομάδες της κοινωνίας. Πρόκειται και για προϊόντα και υπηρεσίες που προϋπάρχουν ή που τώρα αναπτύσσονται. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι φορείς και ομάδες να ξέρουν κατά πόσο μπορούν να έχουν πρόσβαση, πλήρη πρόσβαση σε αυτά τα αγαθά και υπηρεσίες, όπως στην περίπτωση των ε, ιατρικών σκευασμάτων, των φαρμακευτικών σκευασμάτων. Για τους ε, μη βλέποντες θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση και των τυφλών στα φάρμακα διαδικτυακά. Άρα οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι προσβάσιμες για όλους τους ενδυνάμει χρήστες. Το κείμενο αφορά 100 σελίδες και θα ήθελα να διαπραγματευτώ συγκεκριμένες τροπολογίες για να συμφωνήσουμε με τους σκιώδεις και να μπορέσουμε να βρούμε κοινέ λύσεις. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που εκκρεμούν και εγώ δεν είμαι μάγος, θα πρέπει να εργαστούμε συλλογικά και άλλες εμπλεκόμενες επιτροπές να δράσουν. Πρόκειται για μια πολύ πολυσχηδή νομοθετική διαδικασία και θα ήθελα να προωθήσουμε αυτή τη συλλογική εργασία στο μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Kosa. Σας ευχαριστώ κύριε Κόσα. Σκιώδης, ε, από την πολιτική ε, ομάδα ε, S&D είναι η κυρία που δεν είναι παρούσα. Μου ζήτησε όμως ε, να αναγνώσω ένα κείμενο που περιέχει τις πρώτες της αντιδράσεις και φυσικά ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι παρούσα στην σημερινή παρουσίαση του θέματος. Ευχαριστεί τον εισηγητή όμως, τον κύριο Κώσα, για την πολύ πλήρη γνωμοδότησή του. Ωστόσο, επειδή η γνωμοδότηση αυτή ε, ήταν διαθέσιμη μόλις από την προηγούμενη εβδομάδα και περιλαμβάνει τόσο πολλές τροπολογίες, δεν ε, μπορεί να απαντήσει αναλυτικά στις προτάσεις του εισηγητή ε, αυτή τη στιγμή. Η κυρία Πλυνκεβισούτε γενικά είναι της άποψης ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι επικροτέα και την περιμέναμε πολύ καιρό. Ε, πιθανότατα να καταλήξουμε σε ισχυρή νομοθεσία που θα αλλάξει την ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων με αναπηρία καθώς και ηλικιωμένων και άλλων χρηστών στην Ευρώπη, επιτρέποντάς τους πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες ε, με ίσους όρους ε, με άλλους ανθρώπους. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ε, η πράξη για την προσβασιμότητα θα ωφελήσει όχι μόνο τους ανθρώπους με αναπηρία, αλλά και μια πολύ ευρύτερη ομάδα πιο ηλικιωμένων που μάλιστα θα αυξηθεί πολύ τα επόμενα χρόνια. Μια γενική παρατήρηση για το πεδίο εφαρμογής της προτινόμενης οδηγίας. Πρέπει να φροντίσουμε κατά την εργασία μας επάνω στην προτινόμενη οδηγία να θυμόμαστε ότι το πεδίο εφαρμογή ε, προβλέπεται να καλύψει όλου του τομείς όπου υπάρχει ή όπου είναι ε, πιθανό να υπάρξει κατακαιρματισμό της αγοράς. Ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να παρέχεται ένα σωστό περιβάλλον για την παροχή υπηρεσιών και αγαθών, διότι αλλιώς το περιορισμένο πεδίο εφαρμογή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα οδηγήσει ε, στη διαθεσιμότητα κάποιων αγαθών και υπηρεσιών ε, και όχι άλλων. Μάλλον όπου ε, τμήματα μιας υπηρεσίας θα διατίθενται και άλλα τμήματα όχι, που σημαίνει ότι το σύνολο τη υπηρεσία δεν θα είναι προσβάσιμο. Επίσης, συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα άτομα με αναπηρία ε, που θεωρεί ότι το να παρέχουμε προσβασιμότητα δεν αποτελεί εμπόδιο, είναι τρόπος να εξαλείψουμε εμπόδια στη κοινωνία μας ε, και είναι απαραίτητη προϋπόθεση ε, για να απολαύσει κανείς άλλα θεμελιώδη δικαιώματα όπως είναι η πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση, στις δημόσιες υπηρεσίες, την ελεύθερη κινητικότητα κλπ. Για το λόγο αυτό, η προσβασιμότητα ωφελεί όλους τους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των καινοτόμων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων με εταιρική κοινωνική ευθύνη. Γι' αυτό η κυρία Πλινκεβισιούτε προσβλέπει στην εργασία πάνω σε αυτό το σημαντικό νομοθέτημα. Προσβλέπει στην συνεργασία με τον εισηγητή και τους άλλους σκιώδες εισηγητές. Αυτό αυτή... Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις της σκιώδους συγγήτριας της κυρίας Μπλίνκεβισιούτε. Θα δώσω το λόγο τώρα στην επόμενη σκιώδη εισηγήτρια, την κυρία Χέλγα Στίβενς. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Eh, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. να ευχαριστήσω καταρχάς τον συνάδελφό μου, τον κύριο Άνταμ Κόσα, για όλη τη δουλειά που έχει κάνει πάνω στη γνωμοδότηση αυτή. Ο νόμος περί προσβασιμότητας είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία ε, για την ε, εφαρμογή της ε, συνθήκης για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία. Μια συνθήκη που έχει επικυρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για να διασφαλίσει την προσβασιμότητα από όλους σε αγαθά και υπηρεσίες. Στηρίζω την ευρεία προσέγγιση του κυρίου Κώσα όσον αφορά την ομάδα στόχο. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή ποιος θα ωφεληθεί από την νομοθεσία αυτή δεν καλύπτει μόνο ανθρώπους με αναπηρία, καλύπτει όλους. Και γι' αυτό ονομάζεται η νομοθεσία περί ε, προσβασιμότητας ε, και όχι περί ατόμων με αναπηρία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, μια αλλαγή στη νοοτροπία. Η ε, προσβασιμότητα θα ωφελήσει όλους τους πολίτες ε, και όχι μόνο αυτούς με λειτουργικούς περιορισμούς ή με αναπηρία. Θα πρέπει να αναφέρουμε λοιπόν και τους ηλικιωμένους σε μια ομάδα που όλο ένα αυξάνεται και που θα αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Επικροτώ το γεγονός ότι αναφέρεται ο ε, συνολικός σχεδιασμός ε, είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται στον τομέα της πληροφορικής εδώ και πολλά χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε όσο γίνεται περισσότερες υπηρεσίες ε, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Γενικά είμαι υπέρ μιας λειτουργικής προσέγγισης που επιτρέπει χώρο στην καινοτομία, διασφαλίζει ταυτόχρονα πλήρη προσβασιμότητα για όλους. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η καλύτερη προσέγγιση είναι μια υβριδική προσέγγιση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποια πρότυπα όπως αυτά που έχουμε στην οδηγία για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο. Ο ίστατος στόχος άλλωστε είναι η προσβασιμότητα. Προς αυτό το στόχο θα πρέπει να εργαστούμε, αλλά δεν μπορούμε εμείς ως ευρωβουλευτές να ε, υπαγορεύσουμε πώς θα γίνει αυτό. Ο νόμος αυτός θα τεθεί σε ισχύ σε κάποια χρόνια και δεν γνωρίζουμε πόσο γρήγορα οι τεχνολογικές ε, αλλαγές ε, θα, γίνουν. Μπορεί πολύ γρήγορα κάποια πρότυπα να ε, αποδειχθούν ξεπερασμένα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας το θέμα αυτό. Θα πρέπει να φροντίσουμε ακόμα και τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ωφεληθούν από την πιο πρόσφατη τεχνογνωσία. Η ε, καινοτομία και η προσβασιμότητα μπορούν ε, να συνδυαστούν. Δεν αποκλείουν η μία την άλλη και ελπίζω η συνεργασία μας να είναι επικοδομητική και να ωφελήσει όλους τους πολίτες συμπεριλαμβανομένων των πολιτών με αναπηρία. Φυσικά θα είμαι σε επαφή με ενώσεις ατόμων με αναπηρία για να ακούσω τις δικές του απόψεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Μαριαν Χάρκιν είναι η επόμενη σκιώδη συζυγήτρια. Ζητεί συγγνώμη για την απουσία της σήμερα. Και θα στείλει γραπτό στις παρατηρήσεις της ε, στον εισηγητή τον κύριο Κόσα, Διότι δεν υπήρχε συνάδελφος που να μπορεί να την αντικαταστήσει σήμερα. Κάτι που σημαίνει ότι προχωράμε στην κυρία Κούνεβα, που είναι η επόμενη σκιώδη εισηγήτρια και εκπροσωπεί την ΚΟΕ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί και αγαπητέ συνάδελφοι, συγχαίρω καταρχά τον κύριο Κόζα για την γνωμοδότησή του. Χαίρομαι που έχουμε σε πολλά σημεία τις ίδιες απόψεις με αυτές που έχω προσθέσει και εγώ στην γνωμοδότηση που έχω ετοιμάσει για την Επιτροπή Αναφορών. Είμαστε πολύ κοντά στο θέμα του ορισμού, γιατί και εκείνος όπως και εγώ υιοθετεί έναν ορισμό που δεν ρίχνει το βάρος στους ανθρώπους με κάποιους μορφής αναπηρία για την δύσκολη πρόσβαση που έχουν στα προϊόντα, αλλά και θυμίζει πως το περιβάλλον δημιουργεί αυτές τις δυσκολίες. Αναφερόμαστε σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με βλάβες σχετιζόμενες με την ηλικία ή με οποιοδήποτε άλλο ηθείο. Είμαστε επίσης πολύ κοντά στις τεχνικές προδιαγραφές που ζητάμε ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες να είναι πραγματικά προσβάσιμες. Νομίζω πως η γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης είναι πολύ σημαντική και έναν ακόμα λόγο, διότι συνδυάζει εκτός από τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία και ένα ακόμη θεμελιώδες δικαιώμα, το δικαιώμα συνεργασία. Τόσα ζητούμε με αυτή την έκθεση και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις είναι πολύ σημαντικά, διότι διευκολύνοντας τις ζωές των ανθρώπων μπορούμε να δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας. Χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για να βοηθήσει τόσο τους κατασκευαστές να δημιουργήσουν τις προδιαγραφές που χρειάζεται για τα προϊόντα, όσο και τις εταιρείε προ, αλλά και τις εταιρείε δια, διάθεσης των προϊόντων θα κάνουμε κάποιες τροπολογίες προς αυτήν την κατεύθυνση και είμαστε σίγουροι πως θα βρουν την καλή αποδοχή από την εισηγητή. Σε ευχαριστώ πολύ. Thank you. Uh, ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος από τους πρασίνους η κυρία Τζέ έχει το λόγο από το EFTD. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κώσα για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων που έχει μεγάλη σημασία για να δημιουργήσουμε μία βάση διαπραγματεύσεων για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για ένα ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος. Η νέα αυτή οδηγία θα πρέπει να έχει βασικό στόχο την εναρμόνιση των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών, έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να πραγματοποιήσουν τους στόχους και τις εθνικές συμφωνίες με βάση τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ ως προς την προσβασιμότητα σε αγαθά και υπηρεσίες. Αγαθά και υπηρεσίες ε, που διαφέρουν μεταξύ τους. Μιλάμε για τραπεζικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μεταφορών, bankomat ε, και ούτω καθεξής. Άρα το πεδίο δράσης αυτής της οδηγίας είναι ευρύτατο δεν θα πρέπει να συγχέουμε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης της ΙΜΚΟ με την εργασία που έχει γίνει από τη συνάδελφο Στίβενς για τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ε, Εχόντων Αναπηρίες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μία σωστή προσέγγιση και να κινηθούμε προς συμφέρον των ανθρώπων με αναπηρίες και όπως υπενθυμίσαμε πρόκειται για μία ευρύτατη κατηγορία, αφορά και τους γυρεότερους γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη γύρανση του πληθυσμού. Εγώ δεν θα ήθελα να επικρίνω αυτό το πλαίσιο, απλώς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε κοινέ λύσεις με βάση το άρθρο 3 παράγραφος 10. Τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν ως προς τους όρους προσβασιμότητας που ορίζει η οδηγία. Αυτό τι σημαίνει ότι από μία πλευρά η οδηγία θέλει να διευκολύνει την προσβασιμότητα στα αγαθά και υπηρεσίες, όμως τα μέτρα που προβλέπονται δεν είναι δεσμευτικού χαρακτήρα, έτσι ώστε οι άνθρωποι με αναπηρίες να έχουν πλήρη προσβασιμότητα στα αγαθά και στις υπηρεσίες. Στην χώρα μου βλέπω πω ότι υπάρχουν πολλά προσκόμματα προς αυτή την κατεύθυνση γι' αυτό. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα πλαίσιο το οποίο δεν μπορούμε να διαχειριστούμε εύκολα. Αναρωτώ με τι σκέφτεται ο συνάδελφος Κώσα σε σχέση με αυτές τις διατάξεις και κατά πόσο δεν θα ήταν σκόπιμο κατά κάποιο τρόπο να προβούμε σε μία πρόταση πιο δεσμευτική. γιατί έχει σημασία να δούμε και το περιβάλλον αυτών των της παραγωγής αυτής της προσβασιμότητας, της δημιουργίας αυτής της προσβασιμότητας. Το θέμα είναι ύψης της σημασίας. Χτες στην Ιταλία έγινε το δημοψήφισμα για τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και πολύ συχνά βλέπουμε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει πλήρης εποπτεία του πλαισίου παροχών προς τον πολίτη. Μιλάμε και για το δικαίωμα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος. Πολλές φορές είναι δύσκολο. Δεν υπάρχει πλήρης προσβασιμότητα. Σήμερα στην Ιταλία υπάρχουν πολλά σχολεία που είναι εκλογικά κέντρα, τα οποία όμως δεν είναι προσβάσιμα για τα αμαία. Τον Ιούλιο το Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση Stevens με θετικά αποτελέσματα και ήδη αναγνωρίσαμε τη σημασία της καθολικής προσβασιμότητας σε όλες τις κατασκευές. Νομίζω λοιπόν ότι αυτές οι διατάξεις θα πρέπει να εμπεριέχονται και στην πρόταση νομοθετικού περιεχομένου που τώρα συζητείται στην ε, ΙΜΚΟ και θα πρέπει να είμαστε σαφείς ε, όσον αφορά και την Επιτροπή Απασχόλησης. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Κώσα και τους ε, σκιώδεις. Ελπίζω η εργασία να είναι πολύ καλή προοπτικά. Ευχαριστώ πολύ. Ζωέλ Μελέ. Ο κύριος Μαρτέν θα λάβει το λόγο. Εξ ονόματος κυρίας Μελέ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κώσα και την κυρία Στίβενς για αυτό το θέμα, το σοβαρό θέμα των ε, αναπηρίων. Με την οδηγία θέλουμε να βελτιώσουμε την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς έτσι ώστε να αρθούν τα προσκόμματα στην ελεύθερη κυκλοφορία και να διευκολύνουμε την προσβασιμότητα όλων ε, στην κοινωνία. Να μπορούν δηλαδή και οι άνθρωποι με αναπηρίες να κινηθούν αυτόνομα. Αυτό δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και τα κράτη και τις τοπικές αρχές. Και εδώ μιλάμε και για τον δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα για το δημόσιο τομέα. Έχουμε την εντύπωση ότι το θέμα των αναπηριών έχει χειραγωγηθεί υπέρ της εσωτερικής αγοράς για να υπάρξει δηλαδή εναρμόνιση της νομοθεσίας και ενοποίηση της αγοράς. η αυτή την ε, έννοια, αυτή η επικάλυψη οδηγεί σε μία σύγχυση σε σχέση με τις φυσικές δηλαδή αναπηρίες περισσότερο η κύρωση της ε, Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα ΑΜΕΑ αποτελεί, ε, θα πρέπει να ε, θεωρηθεί ως ένα πρόσκομα, δηλαδή είναι ένας δούριος ύπος στην ουσία για να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη ομοσπονδιακού χαρακτήρα. Χαίρομαι γιατί η κυρία Μωρέν Σάρτ και Κοσμήτορας είναι εδώ για να με ακούσει. Η προσβασιμότητα των ανθρώπων με αναπηρία μας απασχόλησε ε, από τον ε, Αύγουστο του 2006 και ιδιαίτερα εμένα γιατί πλέον είμαι μονόφθαλμος γιατί υπέστην μία επίθεση και έχασα το ένα μου μάτι. Και εδώ δεν μιλώ μόνο για το αισθητικό σκέλος. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη το άρθρο 30 έτσι ώστε να μπορέσω εγώ να μεταβώ στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο γιατί δεν μπορώ να οδηγήσω για να μεταβώ στο αεροδρόμιο ή στο σιδηροδρομικό σταθμό. Σε πρώτη φάση λοιπόν οι κοσμήτορες το αρνήθηκαν γιατί μου είπαν ότι όχι, δεν είναι τόσο σίγουροι ότι είμαι πραγματικά μονόφθαλμος και μου ζήτησαν το θέμα αυτό να συζητηθεί από τους πρόεδρους, δηλαδή από τη διάσκεψη των πρόεδρων. Γι' αυτό θα ήταν καλύτερα να ε, ασχοληθείτε με το ίδιο σας το σώμα σε πρώτη ε, φάση και τις ε, αμέλειες που υπάρχουν εκεί. Σας ευχαριστώ. Ίσως η κυρία Μωρέ Σαρτιέ θα μπορούσε να αντιδράσει και να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω την εργασία του συναδέλφου Κόσα και τη συνεισφορά και της κυρίας Στίβενς. Προσδίδω μεγάλη σημασία σε αυτή την εργασία και είμαι ιδιαίτερα προσεκτική στις εξελίξεις ως προς την προσβασιμότητα των ανθρώπων με αναπηρίες, προσβασιμότητα σε όλες τις υπηρεσίες στα κράτη-μέλη. Ως προς τη συγκεκριμένη περίπτωση θα ήθελα να πω ότι ως ε, κοσμήτορας ίσως να μην γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος ότι συνεδριάσαμε με βάση όλα, με τη συμμετοχή όλων των πολιτών με αναπηρίες, των μελών δηλαδή, για να δούμε πώς μπορούμε, των μελών του Κοινοβουλίου, για να δούμε πόσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ε, προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε όλες τις βελτιώσεις για τη συμμετοχή των ε, μελών στις εργασίες μας. Όσο αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, πράγματι το σώμα των κοσμητόρων συνεδρίασε. Έχουμε να κάνουμε με μία μόνιμη ε, αναπηρία ενδεχομένως, γιατί πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι προσωρινή μία αναπηρία ή μόνιμη. Έχει μεγάλη σημασία από όσο καταλαβαίνω, ε, τα όσα προείπε το μέλος, Ε, φαίνεται ότι η αναπηρία θα μετατραπεί σε μόνιμη. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνει νέα αίτηση στο σώμα των κοσμητόρων. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια των προέδρων της, ε, των ομάδων. Εν πάση περιπτώσει το θέμα θα ε, μας υποβληθεί και θα ήθελα ο συνάδελφος να λάβει υπόψη αυτή την τάξη πραγμάτων και τους κανόνες που ισχύουν. Ο κύριος Φουντούλης έχει το λόγο. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον συνάδελφο Κόζα και συνάδελφο Στίβενς για την εργασία τους. Αλλά πώς μπορούμε να μιλάμε για προσβασιμότητα σε αγαθά και υπηρεσίες σε μια Ευρώπη που μόνο ενωμένη δεν είναι στα θέματα των ΑΜΕΑ, θα μου πείτε γιατί το λέω αυτό. Απλά σας ενημερώνω πως από σήμερα 85 Ελληνόπουλα, παιδιά με ειδικέ ικανότητες που φοιτούν στο Σικιαρίδιο Ίδρυμα, στο οποίο φυτά και η κόρη μου, παιδί με σύνδρομο Down, δεν έχουν πλέον πρόσβαση στο σχολείο τους. Η εταιρεία η οποία είχε τα σχολικά έχει μείνει απλήρωτη εδώ και πάρα πολλούς μήνες και έτσι σταμάτησε τα δρομολόγια. Οι γονείς έχουν τεράστιο πρόβλημα γιατί δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά στο σχολείο κάποιοι πρέπει να πάνε στην εργασία τους, ούτε το ωράριο της εργασίας τους ταυτίζεται με το ωράριο του σχολείου. Σε αυτό το σχολείο τα παιδιά αποκτούν νέες δεξιότητες, είναι στα εργαστήρια, ε, προσπαθεί το κάθε παιδί να ενταχθεί στην αγορά εργασίας και να κοινωνικοποιηθεί και δυστυχώς από σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στο σχολείο. Η, η, κρατική επιχορήγηση στο ελόγο ίδρυμα για φέτος είναι μηδενική. Προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση να παρουσιάσει πλεονάσματα, όπως έχει συμφωνήσει με τους εταίρους, έχει αφήσει με τα άτομα με αναπηρίες το έλεος του Θεού. Οι οικογένειες έχουν έρθει σε απόγνωση, γιατί δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους αυτά που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτονόητα. Κάθε φορά που στην Ελλάδα επιβάλλονται περικοπές, τα εύκολα θύματα είναι τα άτομα με αναπηρίες. Έτσι ετοιμάζονται τώρα περικοπές και στα αναπηρικά επιδόματα. Πλέον τα αμαία στην Ελλάδα είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Κύριε Κόσα, εσείς επιθυμείτε να λάβετε το λόγο για να ολοκληρώσετε την ε, συζήτηση του θέματος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για αυτό το ζήτημα ύψης της σημασίας. Είναι δύσκολο να υπάρχει πλήρης κατανόηση του ζητήματος και εγώ αντιμετωπίζω μεγάλες δυσκολίες να διαβάσω το κείμενο λεπτομεριακά και να λάβω υπόψη τη θέση εφαρμογή αυτών των κανόνων. Υποβλήθηκαν πολλές ερωτήσεις και θα ήθελα να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά. Η πρώτη ήταν περισσότερο μια γενική τοποθέτηση και λιγότερο μια ερώτηση σχετικά με το γεγονός ότι το κείμενό μου δεν περιλαμβάνει όλες, όλα τα αιτήματα που προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών σχετικά με την πρόσβαση σε κτίρια καθώς και σχετικά με το πεδίο εφαρμογής. Όμως είπα από την αρχή ότι κρεμούν ακόμη ορισμένα ερωτήματα. Θα συνεχίσω τις διαβουλεύσεις με τους γεωδησιητές, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα με κοινή προσπάθεια, διότι πρόκειται για θέματα που δεν αφορούν βεβαίως τις προσωπικές απόψεις του εισηγητού, ο οποίος έρχεται και ζητεί την υποστήριξη των συναδέλφων του. Πρόκειται για θέματα τα οποία επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή και η λύση τους μπορεί να διευκολύνει τη ζωή μας στο επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι μια πενταετία. Πρόκειται για πρόσβαση σε υπηρεσίες που μας αφορούν όλους. <clears throat> Δέχτηκα και μια ερώτηση για την πρόσβαση στα κτίρια. Θα ήθελα, όχι τόσο για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, ωστόσο να προβάλλω το επιχείρημα ότι πρόκειται για εθνική αρμοδιότητα. Εμείς δηλαδή το λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός αυτό στην εργασία μας. Και λόγω της σταθερής στάσης της Επιτροπής μας, Άρα λοιπόν σε αυτή τη στάση εμείς επιμένουμε πάντοτε να διευκολύνεται η πρόσβαση στα κτίρια όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διαφθορτικά ταμεία εάν στα κτίρια στο εθνικό επίπεδο δεν προσφέρεται επαρκής πρόσβαση. Το πρόβλημα βέβαια αφορά κυρίως κτίρια τα οποία ήδη υπάρχουν παλαιότερα δηλαδή. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά την γύρανση της κοινωνίας. Εγώ συμφωνώ η οδηγία θα αφορά όλο και περισσότερα πρόσωπα. Αλλά, προσοχή, η μεγάλη ηλικία δεν είναι αναπηρία. Υπάρχουν βέβαια όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λειτουργικά προβλήματα. Και επομένως έχουν περιορισμούς στις διάφορες λειτουργίες τους. Και γι' αυτό προτείνω μια λειτουργική προσέγγιση. Θα πρέπει, ωστόσο, να, είναι, να έχουμε υπόψη μας ποιες λειτουργίες θα πρέπει να διασφαλίζει η σχετική υπηρεσία. Δεν θα πρέπει τώρα να συγχαίουμε την ασθένεια με την αναπηρία. Πρόκειται για διαφορετικά πράγματα και γι' αυτό χρειάζεται διακριτή μεταχείριση. Άλλωστε και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι ξεκάθαρη από αυτού. Το 2005 εκδόθηκε απόφαση που ορίζει ότι η πρόσβαση δεν είναι το ίδιο σε περίπτωση ασθένειας και σε περίπτωση αναπηρίας και γι' αυτό πρέπει να ε, υπάρχει διαφορετική μεταχείριση. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, άκουσα τις παρατηρήσεις σχετικά με την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας αυτής για το γεγονός δηλαδή ότι τα παιδιά δεν μπορούν πλέον να πάνε στο σχολείο τους. Δυστυχώς η οδηγία δεν αφορά τέτοια περιστατικά. Πρόκειται για την οδηγία για πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες. Το πρόβλημα που σημειώνει ο συναδελφός μου είναι βαρύτατο και θα πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με αυτό. Εγώ μάλιστα προσωπικά ο ίδιος σημειώνω ότι τα κράτη δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν οικονομίες, να κάνουν περικοπές δηλαδή, σε βάρος ανάπηρων παιδιών. Διότι η πρόσβαση στην παιδεία και στην εκπαίδευση δεν επιτρέπεται να περιορίζεται. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον ε, κύριο εκπρόσωπο του Εθνικού Μετόπου. Δεν νομίζω ότι κάνουμε προσπάθεια να κάνουμε μια ομοιόμορφη αγορά ε, μέσω της οδηγίας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ είναι τα πρόσωπα τα οποία έχουν κάποια αναπηρία και εν πάση περιπτώσει και κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να την χάνει της ισότιμης μεταχείρισης ό,τι αφορά την πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες. Και ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για κάποιον Ούγγρο, Γάλλο, Βέλγο, ο οποίος έχει κάποια αναπηρία, διότι το πρόσωπο αυτό έχει τις ίδιες ανάγκες. Όλα τα πρόσωπα αυτά έχουν τις ίδιες ανάγκες εφόσον έχουν τις ίδιες αναπηρίες. Δεν μιλούμε για ενιοποίηση της αγοράς. Εμείς θέλουμε να είναι ομοιόμορφη, να είναι η πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες. Νομίζω πάντως ότι δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες αποκλήσεις μεταξύ μας, μεταξύ των απόψεών μας. Αυτό που θα είναι πιο δύσκολο θα είναι να καταλήξουμε στις κατάλληλες διατυπώσεις ώστε να συμφωνήσουμε. Θεωρώ πάντως ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Δεν έχουμε βέβαια και πολύ χρόνο. Η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών έχει πολύ περιορισμένο χρονοδιάγραμμα και αυτό αναγκάζει και εμάς να εργαστούμε γρήγορα. Ήδη τούτη την εβδομάδα θα οργανώσω μια συνάντηση με τους κοιόδης και θα κάνω κάθε δυνατή προσπάθεια για να δώσω, ε, τελική μορφή μάλλον στο κείμενό μου όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και Κώσσα. Από την, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν θέλετε μπορείτε να μιλήσετε. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ευχαριστώ βεβαίως τον Ευρωβουλευτή σας κύριο Κώσα που ε, έχει καταθέσει τόσο λεπτομερή γνωμοδότηση και η οποία περιέχει μάλιστα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, ιδίω για το παράρτημα 1, τις λειτουργικές δηλαδή απαιτήσει. Εκεί βλέπει τα πράγματα διαφορετικά από την, από, την πρότασή μας και νομίζω ότι πρόκειται για ουσιώδη συζήτηση σε ό,τι αφορά δηλαδή, το πεδίο εφαρμογή της προτάσεως που θα έχει σχέση με το πώς διαμορφώνεται η πρόσβαση. Εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση που εμάς πάντως μας φαινόταν πιο γενική και πιο ευέλικτη. Ο κύριος Κώσα έρχεται σε απαιτήσει πρόσβασης που είναι αρκετά διαφορετικές. Νομίζω πάντως ότι υπάρχει αντικείμενο συζητήσεως για να μπορέσουμε να βρούμε, να καταλήξουμε στις πιο χρήσιμες επιλογές που να διευκολύνουν και τη βιομηχανία. Για πρώτη φορά πάντως βλέπω τέτοια εργασία προβληματισμού και επανεξέτασης του παραρτήματος που όπως είπα για μένα ανοίγει ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο συζητήσεων. Εξάλλου έχουμε ορισμένα ε, ελάσσονα θέματα, ίσως ερωτηματικά, για ορισμένες τροπολογίες. Πρώτα για τις τροπολογίες που στοχεύουν στην αλλαγή του ορισμού των αναπήρων και των ε, προσώπων με περιορισμένη κινητικότητα. Εμεί κάνουμε μια διάκριση στην πρότασή μας, ώστε να κρατήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τον ορισμό των Ηνωμένων Εθνών. Να έχουμε και έναν ορισμό για τα πρόσωπα με περιορισμένη κινητικότητα. Βάζουμε και τους δύο ορισμούς, βέβαια, όσο μπορούμε εκ παραλίλου, για να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στα, ε, στα ανάπηρα πρόσωπα, το οποίο θα διευκολύνει βέβαια και αυτούς που έχουν περιορισμένη κινητικότητα. Αυτό είναι προφανές. Πάντως κυρίως ο στόχος μας είναι η διευκόλυνση των αναπήρων. Τώρα έχουμε κάποιους δισταγμούς σε ό,τι αφορά ορισμένα σημεία του κειμένου που μας φαίνονται να μειώνουν την υποχρέωση που απορρέει από το Accessibility Act ιδίως τροπολογία 13 για την έννοια της βελτιστοποίησης που για μας σημαίνει μείωση των υποχρεώσεων των κατασκευαστών. Επίσης τροπολογία 39 που επιτρέπει μια στιγμή να το διαβάσω γιατί είναι στα αγγλικά βέβαια οι κατασκευαστές μπορούν να αποφασίσουν να εκτελούν τις απαιτήσει για περιφερειακές συσκευές, για hardware κλπ. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα μπορεί τα ίδια να μην είναι προσβάσιμα, αυτή στιγμή όμως είναι ε, προσαρμοσμένα σε εξωτερικά στοιχεία τα οποία θα τα καθιστούν προσβάσιμα. Αυτό όμως εμεί διαβλέπουμε ότι εδώ υπάρχει ο κίνδυνο να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογή τη προτάσεώ μα. Τέλο δύο ή μάλλον μία αλλαγή που κάπω να το πω, δυσκολεύει, διότι θα έχει σημαντικέ επιπτώσει. Μιλώ για την τροπολογία 26, καθώ επίση και τι τροπολογίε 49 και 60, όπου, όπου εκεί η foreseeable use, η προβλεπόμενη χρήση αλλάζει από τι τροπολογίε αυτές και γίνεται intended use, αυτή δηλαδή η χρήση η οποία, την οποία έχει πρόθεση ο κατασκευαστής να προσφέρει. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, ένα τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο, έτσι, ε, η πρόθεση είναι να μπορεί κανείς να ακούει και να μιλεί. Άρα είναι απολύτως μη προσβάσιμο σε έναν κοφάλαλο. Ενώ αν βάλουμε τη λέξη προβλέψιμη χρήση, foreseeable use, είναι να μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Μέσω αυτού, για παράδειγμα, έχουν γίνει τα διάφορα FE, ε, τηλέφωνα, smartphone και iPhone κτλ. έχουν γίνει πολύ πιο προσβάσιμα, διότι δεν περιορίζονται μονάχα στην ε, φωνητική επικοινωνία. Η προσπάθεια λοιπόν είναι να γίνουν όσο δυνατόν πιο προσβάσιμα και να ανοίξει ο δρόμος σε καινοτομία. Ενώ το άλλο, από το intended use, μπορεί να σημάνει τελικώς μείωση του πεδίου εφαρμογής της ε, προτάσεως. Αυτά είναι τα θέματα στα οποία ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας. Βεβαίως είμαστε στη διάθεση του κ. Κώσα για να συζητήσουμε οποιοδήποτε άλλο θέμα θα ήθελε ή που μπορεί να του φαίνεται χρήσιμο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 11η Ιανουαρίου Εξέταση των τροπολογιών 27 με 28 Φεβρουαρίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης 32 ε, με 23 Μαρτίου και ψηφοφορία στην επί ουσίας αρμόδια επιτροπή θα πραγματοποιηθεί επίσης τον Μάρτιο. Προχωράμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα της ένδυσης. Και δίνω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Τζιν Λάμπερτ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να πω ότι πώς να το πω, αναρωτιόμαστε λίγο τι θα πρέπει να κάνουμε το θέμα αυτό. Υποτίθεται ότι συμβάλλουμε στην ε, έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης ε, για την εμβληματική ε, πρωτοβουλία, η οποία όμως δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα από ό,τι γνωρίζω. Από ό,τι έχω καταλάβει, έχει αναβληθεί λίγο στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Επίσης, όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρά αυτά που γράφω στην παράγραφο 4 της γνωμοδότησής μου, και μπορεί αυτό να ε, παραπλανούν λίγο. Η ε, ε, έκθεση αυτή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν λέει τι πρέπει να κάνουμε και πώ και πού θα βρούμε τη χρηματοδότηση κλπ. Μπορούμε λοιπόν είτε να θεωρήσουμε ότι αποτελεί πρόβλημα αυτό, είτε ότι αποτελεί λευκή σελίδα, στην οποία μπορούμε να καταγράψουμε τα θέματα κλειδιά, τα οποία θέλουμε να, συμπεριλαφ... συμπεριληφθούν στην εμβληματική πρόταση. Ε, το, η αφορμή για την ε, έκθεση αυτή είναι η τραγωδία στην Ράνα Πλάζα πριν από περίπου τρία χρόνια στο Ντακάρ του Μπαγκλαντές. Και έκτοτε έχουμε δει ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παρακολουθεί τη συνέχεια που έχει δοθεί στο συμβάν αυτό και έχουμε επίσης ε, την ε, έκθεση του κυρίου Σούστερ καθώς και έκθεση στην Επιτροπή Εμπορίου. Έχουμε λοιπόν διάφορα στοιχεία στα οποία μπορούμε να βασιστούμε. Από την τραγωδία εκείνη και μετά ε, έχουμε δει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργάζεται με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, με την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές πάνω σε Ε, ένα δικαστήριο το οποίο θα εξετάσει ε, τις ε, συνθήκες ασφαλείας στα κτίρια του τομέα ένδυσης. Επίσης, ο Καναδάς έχει ένα σύμφωνο βιωσιμότητας που αποτελεί μια μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία για να βελτιωθούν οι συνθήκες των εργαζομένων στον τομέα της ένδυσης και ιδιαίτερα στο Παγκλαντές. Η κυρία Ιουγγέριος, ε, αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας ε, και εγώ βρεθήκαμε πρόσφατα στο Παγκλατέ μαζί με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου για να εξετάσουμε τι έχει γίνει στο μεταξύ στον τομέα της ένδυσης, όπου είναι σαφές ότι υπάρχει κάποια βελτίωση όσον αφορά την ασφάλεια των κτηρίων. Ε, τύχθηκαν όμως και διάφορα άλλα θέματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εμβληματική πρωτοβουλία που θέλει να προτείνει οργάνωσε μεγάλη διάσκεψη φέτος στις Βρυξέλλες, ε, όπου συμμετείχαν διάφοροι ενδιαφερόμενοι και όπου εξετάστηκαν τα αποτελέσματα ερευνών εμπειρογνωμόνων που εξετάζουν ε, τον τομέα ένδυσης γενικότερα, όχι μόνο στον Μπαγκλαντές. Ο τομέας της ένδυσης αποτελεί σημαντικό τομέα απασχόλησης, ιδιαίτερα απασχόλησης γυναικών σε πολλές χώρες και ιδιαίτερα στην ε, Νότια ανατολικη Ασία, ακόμα και σε μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είδαμε αλλαγές μετατροπές στον τομέα αυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε λοιπόν ότι σε μια τέτοια πρωτοβουλία θα ήθελε να έχει καλύτερο συντονισμό, καλύτερη συνεργασία, διάλογο, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων, να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εκμεταλλευτεί την προστιθέμενη αξία της Ευρώπης, ε, πιέζοντας όλους τους παράγοντες ε, να ε, εντείνουν τις προσπάθειες για να φροντίσουν να υπάρξει η σωστή ανάπτυξη στις χώρες αυτές και σωστή παγκόσμια διακυβέρνηση. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας επικεντρώνεται στη θέση των ε, απασχολούμενων και όχι τόσο πολύ στον τομέα στο σύνολό του. Και αναφέροντας κάποια πράγματα τα οποία προέκυψαν από τη διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και που μας έχουν πήγει διάφορες ομάδες ε, συμφερόντων. Εντός της ε, αλυσίδας προμήθειας λοιπόν αυτό που αναζητούν διάφοροι είναι διαφάνεια. Δηλαδή να γνωρίζει κανείς ότι όταν αγοράζει κάτι ένα προϊόν του τομέα ένδυσης δεν είναι εις βάρος των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την παραγωγή και ότι ο κατασκευαστής ε, λαμβάνει δίκαιο αντίτιμο καθώς και πληρώνει ε, δίκαιη αμοιβή στους εργαζόμενους του και ότι δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν σημαντικό θέμα όπως και το εισόδημα των εργαζομένων καθώς και τα εργασιακά τους δικαιώματα τα οποία φαίνεται ε, να μην ε, γίνονται σεβαστά σε διάφορες χώρες και μάλιστα με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, κάποιες ε, ζώνες εξαγωγών αποτελούν έχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, οι συλλογικές συμβάσεις, η υγεία και, ο και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η αμοιβή των εργαζομένων, θέματα ισότητας των δύο φύλων. και πώς οι γυναίκες που είναι οι περισσότερες ε, απασχολούμενες στον τομέα αυτών ε, μπορούν να προοδεύσουν ε, στο πλαίσιο του τομέα αυτού, καθώς επίσης θέματα διεύθυνσης, οικειοποίησης κλπ. Κάποια λοιπόν από τα θέματα κλειδιά της γνωμοδότησης και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν πολλοί είναι ότι οι προαιρετικές ρυθμίσεις δεν ε, καλύπτουν επαρκώς τα προβλήματα στον τομέα αυτών. Γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις πρωτοβουλίες που ήδη υπάρχουν και να τις συνδυάσουμε για να υπάρχει συνεπής προσέγγιση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν σαφές και κατά τη διάρκεια της διάσκεψης Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αλλού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε θέση ε, να συνδυάσει διάφορε εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες για να ε, μπορέσει να εφαρμόσει ενιαία πρότυπα, να μην έχουμε διάφορα πρότυπα. Κατά την ε, παραγωγή των προϊόντων ένδυσης, ώστε όποιος φοράει ένα ρούχο να μην νιώθει ότι είναι εις βάρος των επασχολούμενων ε, στον τομέα. Δεδομένου όμως ότι δεν έχουμε πολύ συγκεκριμένη πρόταση μπροστά μας, είναι πολύ δύσκολο να υποβάλουμε τροπολογίες για κάτι που δεν υπάρχει. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λάμπερτ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σούλσες και εισηγητή του ΕΛΚ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρία εισηγήτρια, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια, τη συντάκτρια της νομοδότησης για το σχέδιο γνωμοδότησης που μας έχει υποβάλει. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν επιθυμητό να ε, έχουμε ε, προϊόντα ένδυσης στην Ευρώπη, να μπορούμε να αγοράσουμε προϊόντα ένδυσης, τα οποία να τηρούν περιβαλλοντικά, εργασιακά και άλλα πρότυπα. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί κοινό μας στόχο. Ωστόσο γνωρίζουμε πώς έχει η πραγματικότητα και ξέρουμε ότι με πολλούς τρόπους η τιμή παίζει τελικά ρόλο και ότι πολλοί καταναλωτέ στην Ευρώπη δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για τα προϊόντα ένδυσής του. Άλλη πρόκληση που βλέπω είναι ότι οι χώρε παραγωγή για τι οποίε μιλάμε, διότι ξέρουμε ότι σε μεγάλο μέρο ε, τα προϊόντα ένδυσης ε, δεν παράγονται εντό Ευρώπη, αλλά εκτό. Τίθεται λοιπόν το θέμα. Τι μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα, αν μπορούμε να υποχρεώσουμε ε, τις επιχειρήσεις ένδυσης ε, της Ευρώπης ε, να τηρούν τα πρότυπα. Ε, και αυτό τι σημαίνει, η μεταφορά της ε, ευθύνης ε, του κράτους στις ιδιωτικές εταιρείες. Εγώ θα προτιμούσα να υπάρχουν στην Ευρώπη θελοντικές συμμαχίες για τον βιομηχανικό τομέα, ώστε να φροντίσει να λαμβάνουμε καθαρά εντό εισαγωγικών ρούχα. και σε ε, διεθνές επίπεδο, όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε επίπεδο G20, ε, ΟΣΑ κλπ. Έχω τρεις επικρίσεις ερωτήσεις ε, για το σχέδιο γνωμοδότησης. Σε παράγραφος 8, η εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την ανάπτυξη ενός δίκαιου και σταθερού μηχανισμού τιμολόγηση. Δεν ξέρω ακριβώ τι έχει φανταστεί η συντάκτηρια στο θέμα αυτό αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι προβληματικό όσον αφορά τα καρτέλ. Δηλαδή να έχουμε παρέμβαση στο θέμα της τιμολόγησης. Και όπως ήδη είπα, νομίζω ότι πολύ περισσότερα θα πρέπει να γίνουν σε προαιρετική βάση με μηχανισμούς συμμαχίας που θα οδηγήσουν σε σταθεροποίηση της ε, παραγωγής ρούχων. Αυτή λοιπόν είναι η επίκρισή μου ερώτηση για την παραγραφό 8 και για την παραγραφό 9 έχω επίση μια παρατήρηση. Εγώ θα ήμουν ε, πιο επιφυλακτικός ε, όσον αφορά την διαφάνεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Η αλυσίδα εφοδιασμού είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν πιο χρήσιμο να έχουμε ε, δέσμευση από πλευρά των επιχειρήσεων αντί να έχουμε ε, δεσμευτική νομοθεσία. Αυτέ είναι οι παρατηρήσει μου ω και ο ε, για το σχέδιο γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σούλτσε. Σέρτζιο Γκουτιέρες από την πολιτική ομάδα S&D δεν μπόρεσε να είναι παρόν. Μου έχει υποβάλει όμως ένα κείμενο το οποίο θα αναγνώσω. Θέλει να συγχαρεί την Τζιν Λάμπερτ για το εξαιρετικό κείμενο, το οποίο ευθυγραμμίζεται απολύτως ε, με τις ε, προτεραιότητες ε, της ομάδας S&D. Μεταξύ άλλων δηλαδή, το ότι η πρωτοβουλία για την ένδυση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ε, δράσεις πέρα από την ε, συμμόρφωση και θα πρέπει να στηρίζει την ικανότητα δημοσίων αρχών συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης ε, της εργασιακής διοίκησης και των σχετικών αρχών, διασφαλίζοντας το εθνικό δίκαιο να συμβαδίζει με τις ε, συμβάσεις ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Ε, επίσης, όσον αφορά την καθιέρωση μηχανισμών, αυτό να γίνεται σε συνεργασία με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Συμφων... Χαιρόμαστε, γράφει ο κύριος Κουτιέρες, ότι το σχέδιο γνωμοδότησης αναφέρεται στην επικύρωση και εφαρμογή των συμβάσεων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στις κεντρικές ε, συμβάσεις και ιδιαίτερα την 181 για την επιθεώρηση εργασίας ε, εφόσον αυτές οι επιθεωρήσεις αποτελούν κλειδί για τον εντοπισμό προβλημάτων. Επίσης ε, την 182 όσον αφορά το, τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας. Η παιδική εργασία είναι διαβοήτη και θα πρέπει να αποτελέσει μία από τις βασικές προτεραιότητές μας. Επίσης, ε, η Σύμβαση 138 για την ελάχιστη ηλικία απασχόλησης. Ε, επίσης, ε, ισότητα των δύο φύλων. Θα πρέπει αυτή η νομοθεσία ενεργά να προωθεί την ισότητα των δύο φύλων σύμφωνα με τις συνθήκες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας 100 και 111. Ο κύριος Γκουτχέρε, σε συμφωνεί με την παράγραφο 5, θα ήθελε όμως να ενισχυθεί το κείμενο στο σημείο αυτό. Οι δράσεις που θα προκύψουν από την εμβληματική πρωτοβουλία να προωθούν τον ε, κοινωνικό διάλογο και τις ε, συλλογικές διαπραγματεύσεις σε όλα τα επίπεδα. Όπου είναι δυνατόν, εκπρόσωποι των εργαζομένων ε, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην διαδικασία δεουσα επιμέλειας και οι δράσει που αναλαμβάνονται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωση, θα πρέπει να προωθούν ε, την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα με συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, οι συμβάσει του Διεθνού Γραφείου Εργασία, οι κατευθυντήρε γραμμέ ε, του ΟΣΑ, καθώ ε, και οι ρυθμίσει του Διεθνού Γραφείου Εργασία για την αξιοπρεπή εργασία και τι αλυσίδε εφοδιασμού, καθώ και οι δράσει που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο τη εμβληματική πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών όσον αφορά τα προϊόντα που αγοράζουν, όπω αναφέρατε και εσεί η ίδια, κυρία Λάμπερτ. Κλείνει την επιστολή του ο κ. Κουτιέρες, ευχαριστώντας και πάλι την Τζιν για τη σκληρή δουλειά της. Ε, πιστεύουμε ότι το κείμενο αυτό είναι καλό και θα αποτελέσει καλή βάση για συμβιβασμό. Η Γιάννα Σιτνάνσκα είναι η επόμενη σκοιότητα εισηγήτρια. Δεν έχουμε όμως κανένα παρόντα από το ECR, ούτε από την ALDE, ούτε από την GUE, ούτε από το EFTD. Ο κύριος Μαρτέν από το ΙΕΝΕΦ e είναι παρόν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Merci. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κατανοώ όταν η κυρία Λαμπέρ λέει ότι ήταν δύσκολο να γίνει μία γνωμοδότηση. Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί βιώνουμε μία κατάσταση πλήρους καταστροφής και στον τομέα της ένδυσης μεταξύ άλλων. Αλλά ξεχνά τα αίτια. Η παγκοσμιοποίηση και οι πολιτικές, οι παράλογες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυστυχώς εθελοτυφλή η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η παραγωγή στην Ευρώπη όπου οι προδιαγραφές είναι υψηλές. Επίσης, ενώ αρχικά μιλούσαμε για ένα φόρουμ ανταλλαγής καλών πρακτικών, φτάνουμε σε μια νομοθεσία όπως την επιθυμεί το Κοινοβούλιο. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την κυρία Λάμπερτ με ορισμένες προτάσεις ε, τροπολογίας. Να ζητήσουμε από την Επιτροπή να υποβάλει τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας αυτής στο Κοινοβούλιο. Δεύτερον, να υπογραμμίσουμε ότι εν ώψη της παγκοσμιοποίησης ο τομέας της ένδυσης μεταφέρεται σε χώρες με χαμηλούς μισθούς και χαμηλή προστασία οδηγώντας σε μαζικές απολύσεις στην Ευρώπη και την απομάκρυνση του τομέα αυτού από την Ευρώπη. Επίσης, ε, στις δημόσιες προμήθειες θα πρέπει να μιλήσουμε για ένα προτιμησιακό καθεστώς καθώς και την προέλευση των προϊόντων, πληροφόρηση για την προέλευση των προϊόντων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη όλες τις προδιαγραφές ε, παραγωγής, να μην σταθούμε μόνο στις τιμές και να κινηθούμε προς αυτό το τομέα και με τις νομοθεσίες μας, με την νομοθεσία μας. Θα πρέπει όμως να είμαστε πιο επικριτικοί γενικότερα, γιατί πρόκειται για μία πρωτοβουλία Ε, η οποία ε, είναι μία πλήρης υποκρισία, μιλώντας για προστασία και κείμενα τα οποία δεν έχουν καμία χρήση. Μιλάμε για συστάσεις, αισθανόμαστε καλύτερα και ξεχνάμε ότι 1.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Μπαγκλαντές οι Κινέζοι και οι Ινδοί θα συνεχίζουν να εργάζονται κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Και παρόλα αυτά υποστηρίζουμε αυτές τις ε, πολιτικές οι οποίες είναι απαράδεκτες. Η παγκοσμιοποίηση λοιπόν οδηγεί σε παραγωγή από σκλάβους πολύ μακριά από την Ευρώπη για να ε, πουληθούν αυτά τα προϊόντα στους ανέργους μας. Ε, λυπάμαι κυρία Λαμπέρ, ε, είσαστε πολύ θαραλέος άνθρωπος, αλλά θεωρώ ότι αυτό το κείμενο δεν μπορεί να αποδώσει. Ευχαριστώ. Εντάξει. κύριος Κάρουνεν έχει το λόγο και εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, όπως ε, ε, έδειξε και η συζήτηση, ο τομέας είναι ιδιαίτερα περίπλοκος και ήθελα να πω ότι η Ευρώπη δεν αφυπνίζεται τώρα. Έχει γίνει σοβαρή εργασία, είναι γεγονός βεβαίως ότι εργαζόμαστε για να δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η πρωτοβουλία στον τομέα της ένδυσης. Βεβαίως δεν υπάρχει κενό. Εγώ προέρχομαι από την πλευρά της ανάπτυξης, από τη Γενική Διεύθυνση της Ανάπτυξης και πολλοί θα μπορούσαν να σας πούν τα ίδια για αυτή την προσέγγιση. Βεβαίως φέρουμε μεγάλη ευθύνη και πρέπει να βελτιώσουμε τα πράγματα σε αυτό το τομέα. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή και εδώ μιλώ εξ ονόματος της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΒΚΟ είναι να υποστηρίξουμε τις δραστηριότητες μέσω της ε, αναπτυξιακής χρηματοδότησης και προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Φέτος υποστηρίξαμε ένα ταμείο που ασχολείται με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και προσπαθεί να προτρέψει, να αποτρέψει, με συγχωρείτε, ατυχήματα δυνάμει των αποφάσεων των G7 και για να προτείνουμε και σωστές αλλαγές στον τομέα της ε, ένδυσης. Ε, επίσης ένα άλλο παράδειγμα αφορά 95 ε, project με τις ΜΜΕ για να γίνουν πιο πράσινες, ιδιαίτερα στην Ασία. Συμφωνώ επίσης με τα σχόλια που αναφέρουν ότι θα πρέπει να χτίσουμε αυτές τις ικανότητες μέσα στα πλαίσια της αναπτυξιακής προσπάθειας. Μέσα στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας θελήσαμε να συνεχίσουμε αυτή την εργασία με χρηματοδοτική αρρωγή στις χώρες που παράγουν, αλλά να προωθήσουμε και τις βέλτιστες πρακτικές και να διαδώσουμε αυτές τις πρακτικές. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν διαφορετικές ε, αποτιμήσεις και θα πρέπει να φτάσουμε σε κάτι το ευρωπαϊκό, αλλά δεν είναι κάτι το τόσο απλό. Γιατί υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες από πλευράς βιομηχανίας και βεβαίως η ουσία είναι πώς συμπεριφέρονται οι ίδιοι οι καταναλωτές στο τέλος. Γιατί πολλές φορές θέλουν να αγοράσουν ευθυνά προϊόντα που παράγονται υπό επώδυνους και αμφισβητήσιμους όρους. Και γι' αυτό, όπως είπα, προσπαθούμε να δούμε ποια μορφή θα λάβει αυτή η πρωτοβουλία στο τέλος. Ευχαριστώ. Η κυρία Λάμπερτ θέλει να μας πει κάτι καταληκτικά. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και για τα σχόλια. Όταν ε, δούμε τις δικές μας ευθύνες, τις εξετάσουμε, βεβαίως ε, κατανοούμε ε, ότι υπήρχαν πολλές έδρες φτηνού κόστους και μετατοπίσεις και αυτό μπορούμε να το δούμε αν συζητήσουμε ιδιαίτερα με τα κροατικά συνδικάτα. Υπάρχουν δηλαδή προβλήματα και στα ίδια τα κράτη τα μέλη. Θα πρέπει να το ε, αντιμετωπίσουμε με βάση την καθημερινή μας εργασία και σε αυτή την Επιτροπή. Και ένας από τους τρόπους είναι να δούμε τι έγινε στο Μπαγκλαντές, ε, τι γίνεται στο Πακιστάν, στην Καμπότζη, έτσι ώστε να κινηθούμε λίγο γρηγορότερα σε σχέση με τα δικά μας φαντουργικά Δεν μπορούμε να είμαστε συγκαταβατικοί. Έγινε ο λόγος για τις δημόσιες προμήθειες, για το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και επίσης θα πρέπει να δούμε και το κόστος της, ε, των μεταφορών. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς κινούνται αυτές οι συμβάσεις και το είδαμε και στο Λονδίνο αυτό. Μας ενδιαφέρει λοιπόν ε, να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε με βάση την αλυσίδα αξιών. Γνωρίζουμε ότι τα προϊόντα που αγοράζουμε και καταβάλουμε χαμηλό αντίτυπο, ξέρουμε από πού προέρχονται πολλές φορές μπορεί να καταβάλουμε υψηλό αντίτιμο, αλλά οι εργαζόμενοι εργάζονται υπό ε, επώδυνες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, μας ενδιαφέρει αυτή η παγκόσμια τάση των ε, ειδών ε, ένδυσης. Οι τιμές πέφτουν και εάν δείτε τα τζιν που αγοράζετε, Πολλές φορές μείωση τιμών ανέρχεται σε 50% ή θα είναι οι ίδιες ε, τιμές που, με αυτές που ήταν 10 χρόνια πριν και δεν μπορεί να το πει κανείς για πολλά προϊόντα. Άρα το θέμα της τιμολόγησης είναι ουσιώδες και αυτό μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σε σχέση με μια ποσοστία αναλογία που αποδίδεται στους εργαζόμενους. Και αυτό είναι ένα μέρος των συζητήσεων και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στα πλαίσια μιας διάσκεψης. Άρα ενδεχομένως θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα που έθιξε ο κύριος Σούλτσε. Ξέρω ότι υπάρχουν ζητήματα στην Επιτροπή όταν μιλήσουμε για τον ε, δεσμευτικό ή εθελούσιο χαρακτήρα. Είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει στην Επιτροπή και με τους ε, σκιώδεις, κάτι το οποίο πιστεύω θα γίνει νωρίς του χρόνου. Θα πρέπει να δούμε πώς θα προωθήσουμε τις συμμαχίες μας ε, μέσα στα πλαίσια μιας τυποποίησης. Αυτό είναι ύψης της σημασίας και εάν μιλήσετε με τους ε, παραγούς του Μπαγκλαντές θα σας πούν ότι ένα από τα ουσιώδη προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι ότι στην ίδια επιχείρηση ανάλογα με το που βρίσκεται κανείς υπάρχουν διαφορετικές ε, προδιαγραφές ασφαλείας. Και αυτό το βλέπουμε και στις διάφορες επιθεωρήσεις. Ως προς το ΔΟΕ νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς ε, προωθούνται οι γνωμοδοτήσεις του και θα εργαστούμε και σε αυτό το τομέα. Καλωσορίζω τα σχόλια για ενίσχυση αυτών των σημείων με ειδική μνήμα. ως προς τις γενικότερες πολιτικές ίσως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, αλλά η κλωστοϊφαντουργία γνωρίζουμε ότι πάντα ε, έπρεπε να διανύσει τα σύνορα ιδιαίτερα για να βρούμε πρώτες ύλες και πριν φτάσουμε στο τελικό προϊόν. Βεβαίως έχει επιτελεστεί κάποια πρόοδος, αλλά μας ενδιαφέρει να ε, υψώσουμε τον ε, πύχη των προδιαγραφών. Και ε, αν δεν είχε νόημα να κάνουμε κάτι τέτοιο, τότε θα κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά αν δούμε τα αποτελέσματα, υπάρχουν βελτιώσεις. Και αυτό βλέπουμε, το είδαμε και στο Μπαγκλαντές την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι εξαιρετική η κατάσταση, αλλά πολύ καλύτερη από δύο-τρία χρόνια και η Επιτροπή για την Νοτιοανατολική Ασία θα συνεδριάσει την 5η στις 2 όπου θα μιλήσουμε με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας για το τομέα ένδυσης σε πολλές χώρες. Ε, προσβλέπω στις ε, τροπολογίες που θα υποβληθούν από τους συναδέλφους και θα προσπαθήσουμε να ε, συντάξουμε την τελική γνωμοδότηση το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών η 8η Δεκεμβρίου, το μεσημέρι. Η έγκριση 25 με 26 Ιανουαρίου 2017. Στην αρμόδια επιτουσίας επιτροπή θα γίνει η ψηφοφορία 20 με 21 Μαρτίου 2017. Αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη. Και έγκριση ε, στην Ολομέλεια πλέον προβλέπεται για τέλη Απριλίου. Να πάμε τώρα στο υπαριθμό 5 της ημερησίας διατάξεως, λειτουργία του franchising στο λιανικό εμπόριο και ε, δίνω το λόγο στον ε, εισηγητή κ. Ματέμ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω την μεγάλη τιμή να ομιλώ ε, ε, με παρουσία τεσσάρων ή πέντε ευρωβουλευτών, αν μετρήσω και εσάς. Και διερωτώ με τι νόημα έχει αυτό. Ειλικρινά. Τέλος πάντων, θα σας πω τα σχετικά με τη γνωμοδότηση για το franchising, η δικαιόχρηση στα ελληνικά, παρόλο που δεν είμαι η Δήμων, Έχω όμως κάποια εμπειρία διότι ως επαγγελματίας επί μια 20 ετία ήμουν επικεφαλής μιας επιχειρήσεως λιανικού εμπορίου που είχε μεταξύ 20 και 30 υπαλλήλων, ένα κατάστημα δηλαδή, το οποίο είχε και franchising, αφενός παπούτσια της μάρκας Charles Jourdan, που στο μεταξύ όμως έχει πτωχεύσει, και άλλοι εταιρεία, πάλι ε, Γάλλος κατασκευαστής παπουσιών, που επίσης πτώχευσε. Ε, μετά από τα υφαντουργικά, δηλαδή πήρε το ποτάμι και, ε, και το υπόδημα στη Γαλλία. Θα είμαι σύντομος γιατί είπα ότι είμαστε πολύ λίγοι το, αυτό το franchising, η δικαιόχρηση, έδινε το, τη δυνατότητα σε πολλούς να ανοίξουν επιχειρήσεις και μάλιστα να δημιουργήσουν και απασχόληση. Όμως και επειδή έχω διαβάσει την έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής ΙΜΚΟ που φαίνεται να ανησυχεί μήπως και αυτοί που εκχωρούν τα δικαιώματα δικαιόχρησης παραμεγαλώσουν, η επένδυση είναι 100% ε, φορτίζεται δηλαδή με την ε, επένδυση 100% αυτός που αναλαμβάνει, που παίρνει την, ε, το franchising. Και μπορεί να έχει και θηγατρικές που κάνουν την διακόσμηση των καταστημάτων και αυτά τα κάνει αυτός που χωρείται ο δικαίωμα της δικαιοχρήσης. Είναι πολύ διαφορετικές βέβαια νομοθεσίες των χωρών μελών είναι αυτονόητο αυτό. Μετά στην παράγραφό μου 4 ζητώ από τις χώρες μέλη να προστατεύσουν αυτόν που λαμβάνει το δικαίωμα της εκχώρησης έτσι και να λαμβάνουν μέτρα για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Άρα η δικαιόχρηση να γίνεται σε τιμές αγοράς, αυτός που εκχωρεί το δικαίωμα δικαιόχρησης να μην επιβάλλει περιοριστικούς όρους που να οδηγούν στην ασφυξία αυτού που λαμβάνει το δικαίωμα. Η αποκλειστικότητα της μάρκας και των προϊόντων της να είναι εγγυημένε από αυτόν που εκχωρεί το δικαίωμα σε αυτόν που το λαμβάνει. Η τροποποίηση των συμβατικών όρων χωρίς διαβούλευση των δύο μερών να απαγορεύεται, το ίδιο να απαγορεύεται και οποιαδήποτε τροποποίηση των συμβατικών όρων με αναδρομική ισχύ. Να διευκολύνεται ο ρόλος των, ε, αυτών που λαμβάνουν το δικαίωμα δηλαδή της δικαιόχρησης, να εναρμονιστούν οι διατάξεις αυτές μεταξύ των χωρών μελών και τέλος να εκπροσωπηθούν, να βελτιωθεί η εκπροσώπηση στα διάφορα συλλογικά όργανα αυτών που ε, λαμβάνουν το δικαίωμα της δικαιόχρησης. Ευχαρίστω θα συνεργαστώ με τους κοιόδης συγγήτες και ιδίω τον κύριο Κάζα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ε, με την κυρία Στάιν Ρουκ των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και θα εξετάσω τις τροπολογίες που θα υποβάλουν... για να φτάσουμε σε μια συνενετική τοποθέτηση. Εγώ δεν προτείνω τίποτε το επαναστατικό, αλλά θέλω να αποφύγουμε πράγματα τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν, γιατί αυτά υποσκάπτουν τη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ και Μαρτά. Δεν είναι παρόντες σκιώδεις εισηγητές. Και από ό,τι καταλαβαίνω μόνο οι δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες, δηλαδή το Λαϊκό Κόμμα και οι Σοσιαλιστές και οι Δημοκράτες έχουν ορίσει ε, εισηγητές για το θέμα. Ίσως τότε μου επιτρέπετε να δώσω τον λόγο στην νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης δηλαδή, η οποία η εκπρόσωπος είναι η κυρία Φρέριξεν είναι παρούσα. Μπορείτε να εξηγήσετε κάπως την θέση της Κομισιόν για το θέμα. Ορίστε κυρία Φρέριξε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λάβαμε το κείμενό σας κύριε Σιγητά προ δύο ημερών. Το έχουμε λάβει υποσημείωση. Δεν έχουμε όμως ακόμα σχέδιο ψηφίσματος και γι' αυτό δεν έχουμε και εμείς ακόμη τελική θέση για τις προτάσεις σας. Τις εξετάζουμε. Θα επαναλάβω αυτά που είπα και στην Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών, ΙΜΚΟ, ότι για να μπορέσει να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτού χρειαζόμαστε ενδείξεις του διασυνοριακού χαρακτήρα του θέματος. Ότι είναι δηλαδή θέμα το οποίο άπτεται της ενιαίας αγοράς διότι από αυτά που βλέπουμε ως τώρα, αντιλαμβανόμαστε βεβαίως τα προβλήματα που επισημαίνεται ότι υπάρχουν, αλλά αυτά είναι προβλήματα εγχώρια των χωρών μελών. Αυτό που μας χρειάζεται είναι ξεκάθαρες ενδείξεις ότι υπάρχει εδώ διασυνοριακός χαρακτήρας ε, του προβλήματος. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής κατάθεση τροπολογιών μέχρι τις 13, 13 συγγνώμη, 12 Έγκριση στην απασχόληση 23 Φεβρουαρίου. 24-25 στην ΙΜΚΟ και στην Ολομέλεια ακόμη δεν έχουμε ημερομηνία. Ευχαριστώ κύριε Μαρτά. Ε, θα προχωρήσω τώρα στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως. το 6 δηλαδή, μεταρρυθμίσεις της ελληνικής αγοράς εργασίας. Αυτό το έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη. Ίσως τότε που ήταν στο αποκορύφωμά της η κρίση. Τώρα φαίνεται πως κάπως την συνηθίσαμε την κρίση και δεν τη συζητούμε, δεν τη συζητούμε τόσο συχνά όπως τότε που είχε ας πούμε πρωτοαρχίσει. Θα ήθελα πρώτα να σας καλωσορίσω εδώ κύριε Πέδρο Μάρτινς που είστε μέλος των ε, εμπειρογνωμόνων των θεσμών για θέματα κρίση της ελληνικής αγοράς. Είσαστε από την σχολή Queen Mary's Business and Management του ε, Πανεπιστημίου του Λονδίνου και είστε καθηγητής εφαρμοσμένων οικονομικών και έχετε αναμειχθεί στην διαχείριση της κρίσεως. Και ευχαρίστως θα ακούσουμε να μας πείτε πώς βλέπετε τις μεταρρυθμίσεις στην ελληνική αγορά εργασίας. Από τους Έλληνες ευρωβουλευτές κανείς δεν είναι εδώ, λέει η Πρόεδρος. Προφανώς κάνει λάθος. Όμως ε, είναι πρόσωπα τα οποία ενδιαφέρονται πολύ για το θέμα και άλλωστε όλοι και όλες ενδιαφερόμαστε σε αυτή, για αυτή την ελληνική τραγωδία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ μάλλον να σας δώσω το λόγο για να μας προσφέρετε ίσως κάποια ελπίδα. Thank you very much for the, the invitation. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να έρθω εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης και να παρουσιάσω τα ευρήματα της ομάδας επιρροχνομόνων για τις μεταρρυθμίσεις ε, της αγοράς εργασίας ε, στην Ελλάδα. Όπως αναφέρθηκε, είμαι μέλος ε, της ομάδας επιρροχνομόνων που συναντήθηκε αρκετέ αρκετές φορές το περασμένο έτος για να υποβάλει συστάσεις σχετικά με μελλοντικές πιθανές προσαρμογές στους φορείς ε, της ελληνικής ε, αγοράς εργασίας. Όλοι ανησυχούμε ε, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε λόγω της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας και η ομάδα εμπειρογνωμόνων ήθελε να υποβάλει χρήσιμες συστάσεις για να μπορέσουμε να προοδεύσουμε. Από ό,τι κατάλαβα, μια σύντομη εκδοχή και μια πιο αναλυτική εκδοχή των συστάσεων ε, έχει διατεθεί στους ευρωβουλευτές της Επιτροπής σας. Ε, θα σας παρουσιάσω μια σύντομη επισκόπηση κάποιων από τα αποτελέσματα και νομίζω ότι κατόπιν θα υπάρξουν ε, ερωτήσεις και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε. Όσον αφορά Ε, το πλαίσιο. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ε, η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του μνημονίου που υπογράφει τον Αύγουστο του 2015, όπου υπήρχε συγκεκριμένη διάταξη για την ε, διαδικασία διαβούλευσης, όπου θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, συνολικά 8 καθηγητές από διάφορα πανεπιστήμια της Ευρώπης, εμπειρογνώμονες στο τομέα του εργασιακού δικαίου Ε, του σχετικού οικονομικού τομέα κλπ. Τέσσερις φορές συνολικά συναντήθηκε η ομάδα αυτή, κυρίως στην Αθήνα. Είχαμε υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς ε, και από την κυβέρνηση της Ελλάδας. Η ομάδα είχε τη δυνατότητα να συναντηθεί με, διάφορους, ε, με διάφορες ομάδες συμφερόντων στην Ελλάδα ιδιαίτερα συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις εργοδοτών, την ε, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ε, διαμεσολαβητές και συμβουλευτήκαμε και διάφορους εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις προκλήσεις και τις ε, πιθανές απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Φυσικά είναι πολύπλοκο το θέμα. αντικατοπτρίζει διάφορε απόψεις σε διάφορες προοπτικές. Ωστόσο, με ικανοποίηση σημειώνω ότι παρά τη διάσταση απόψεων υπήρχαν διάφοροι τομεί όπου ε, πέτυχαν συνένεση τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Επίσης, υπήρξαν ε, τομεί όπου ήταν ε, πιο πολλωμένε οι απόψεις στις οποίες δεν μπόρεσε να σημειωθεί συνένεση. Επίσης θα ήθελα να σημειώσω ότι όσον αφορά τον στόχο του μνημονίου, Υπήρχε ιδιαίτερο επίκεντρο στις ε, συλλογικές συμβάσεις, ε, τις συλλογικές απολύσεις ε, και τις εργασιακές δράσεις. Στα θέματα αυτά ζητήθηκε από την ομάδα να υποβάλει συστάσεις. Θεωρήθηκε ότι και διάφοροι άλλοι σχετικοί τομείς έχουν σημασία, ιδιαίτερα όσον αφορά τον ελάχιστο μισθό καθώς και των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης. Ε, στις συστάσεις θα ακολουθήσω την ε, ίδια σειρά που θα βρείτε στα έγγραφά σας. Όσον αφορά τις συλλογικές δράσεις, τις συλλογικές κινητοποίησεις, η ομάδα συζήτησε την πιθανή προσαρμογή στους κανόνες για τις απεργίες, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα. Και ένας από τους στόχους της ομάδας ήταν να χρησιμοποιήσει βέλτιστες πρακτικές από άλλα μέρη της Ευρώπης για την μεταρρύθμιση των σχετικών φορέων στην Ευρώπη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ομάδα κατέληξε σε συνένεση. Θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για προσαρμογές όσον αφορά τις διατάξεις για τις απεργίες. Σχετικό θέμα στη σύσταση 2 είχε να κάνει με τα lockouts. Και πάλι η ομάδα θεώρησε ότι ούτε και εδώ υπάρχει ανάγκη για προσαρμογή με βάση βέλτιστες πρακτικές από άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλο θέμα στο οποίο επικεντρώθηκαν ε, οι επιρρογνώμονες είχε να κάνει με τις συλλογικές απολύσεις. Και αυτό είναι ευαίσθητο θέμα, διότι μπορούν να επηρεαστούν τα επίπεδα απασχόλησης από τις διατάξεις που έχουν να κάνουν με τις συλλογικές απολύσεις. Η ομάδα διαπίστωσε τους ε, περιοριστικούς κανόνες και τις περιοριστικές πρακτικές ε, που ισχύουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάγκη για διοικητική έγκριση από το Υπουργείο για να πραγματοποιηθεί η συλλογική απόλυση. Και αυτό εξηγεί τον σχετικά χαμηλό αριθμό τέτοιου τύπου προσαρμογών και μπορεί να παίξει ρόλο σε άλλου τύπου προσαρμογές που μπορεί να αποδειχτούν πιο βλαβερές ε, όσον αφορά την απασχόληση. Ενώ υπήρχαν διαφορές ε, στις απόψει ε, των διαφόρων μελών, γενικά υπήρχε συνένεση ότι κάποια προσαρμογή είναι απαραίτητη. Πιθανότατα είναι απαραίτητη υπομορφή ε, απάλληψης αυτού του κανόνα. Ωστόσο, κάποια μέλη της ομάδας θεώρησαν ότι μάλλον επεσήμαναν ότι το θέμα αυτό εξετάζεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και υπάρχει άποψη του Γενικού Εισαγγελέα, ωστόσο ε, επισημάνθηκε ότι είναι προτιμητέο να περιμένουμε και να ακούσουμε πρώτα τι έχει να πει το δικαστήριο για το συγκεκριμένο θέμα. Όσον αφορά τη σύσταση 4, έχει να κάνει με τη μερική απασχόληση. Γενικά και εδώ υπήρχε συνένεση, μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά ε, την ε, απασχόληση βραχίας διαρκείας. ώστε να μπορούν ε, επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν περιόδους κρίσης, ώστε να μην είναι απαραίτητη πλήρης απόλυση. Δηλαδή, αν ε, μπορεί η επιχείρηση να ε, απασχολεί για σύντομο χρονικό διάστημα κάποιο απασχολούμενος, αυτό θα μπορέσει να βοηθήσει τις επιχείρησεις αυτές σε εποχές κρίσης. Αυτό όμως απαιτεί περισσότερες επενδύσεις από πλευράς της κυβέρνησης όσον αφορά τα επιδόματα ανεργίας για τα διαστήματα ε, όπου ο εργαζόμενος θα καλύπτεται από ένα τέτοιο πρόγραμμα ε, απασχόλησης βραχίας διαρκείας. Επίσης, όσον αφορά τις συλλογικέ ε, διαπραγματεύσεις ε, και τον ελάχιστο μισθό, υπήρχε κάποια διαφωνία ανάμεσα στους εμπειρογνώμονες σχετικά με το ποιος θα είναι ο πιο αρμόδιος για τον καθορισμό του ελάχιστου μισθού, του ελάχιστου εισοδήματος. Κάποια μέλη της ομάδας ε, θεώρησαν ότι θα ήταν προτιμητέο η κυβέρνηση να έχει όλη την ευθύνη στο θέμα αυτό, ενώ άλλα μέλη της ομάδας θεώρησαν ότι θα πρέπει να εναπόκειται στους κοινωνικούς εταίρους τις ε, ενώσεις ε, εργοδοτών και εργαζομένων να αποφασίσουν σχετικά με το κατάλληλο επίπεδο του ε, ελάχιστου μισθού. Αυτό ίσχυε άλλωστε στην Ελλάδα το 2011. Έγιναν όμως σημαντικές αλλαγές και υπάρχει σύσταση η κυβέρνηση να καθορίσει τον ε, ελάχιστο μισθό ε, κατόπιν διαβούλευσης. σχετικό θέμα συζήτησης, όπου δεν καταλήξαμε σε συμφωνία, τα διάφορα μέλη της ομάδας, είχε να κάνει με ε, το, τους ελάχιστους μισθούς, ε, το ελάχιστο ημερομίσιο νέων. Κάποια μέλη της ομάδας ε, θεώρησαν ότι το παρόν σύστημα που καθορίζει το ελάχιστο εισόδημα ανάλογα με την ηλικία του εργαζομένου θα πρέπει να διατηρηθεί, ενώ άλλα μέλη της ομάδας θεώρησαν ότι το ισχύον σύστημα χαμηλότερου ελάχιστου μισθού για τους πιο νέους θα πρέπει να εξαλειφθεί. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και εδώ είχαμε διάφορες ε, συστάσεις. Ε, κάποιες από αυτές ε, βρήκαν συνένεση στην ομάδα, ενώ άλλες όχι. Ένας τομέας όπου υπήρχε συνένεση μεταξύ των μελών της ομάδας είχε να κάνει με τις ε, πρακτικές παράτασης, ε, δηλαδή το αν μια συλλογική σύμβαση μπορεί να καλύπτει όλους τους εργαζομένους ε, ή όλες τις επιχειρήσεις σε έναν συγκεκριμένο τομέα, πέρα από τα μέλη των οργανώσεων που καταλήγουν στη συμφωνία. Υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στο θέμα αυτό. Η ομάδα συμφώνησε ότι θα πρέπει να είναι δυνατόν να μπορεί να διευρυνθεί μια συλλογική σύμβαση εφόσον ε, πληρούνται ένα συγκεκριμένο κριτήριο, ένα συγκεκριμένο ποσοστό ε, των εργαζομένων να εργάζονται σε επιχειρήσεις που συμμετείχαν ε, στις διαπραγματεύσεις. Στις κάτω χώρες, για παράδειγμα, στη Γερμανία, σε κάποιο βαθμό και στην Πορτογαλία ισχύει ένα τέτοιο σύστημα. Και αυτό ήταν και το κριτήριο που ίσχυε στην Ελλάδα μέχρι το 2011. Παρότι αμφισβητήθηκε το αν οι αρχές είχαν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ε, για να διασφαλίσουν την παρακολούθηση του κριτηρίου εκπροσώπησης. Όπως και να έχει, η σύσταση 7 πράγματι δείχνει ότι η εισαγωγή της αρχής της διεύρυνσης ε, με βάση το κριτήριο αυτό θα ε, αποτελέσει σωστή ε, και χρήσιμη μεταρρύθμιση. Ωστόσο, υπήρχαν κάποιες στοιχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων όπου δεν υπήρξε συνένεση στην ομάδα. Για παράδειγμα, το θέμα της το, ε, το θέμα του κατά πόσο ε, συλλογικές διαπραγματεύσεις σε χαμηλό επίπεδο θα υπερισχύουν ε, αυτόν ε, υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή, αν σε επίπεδο τομέα η συμφωνία υπερισχύει της συμφωνίας στην επιχείρηση. Ε, κάποιοι θεωρούν ότι το υψηλό επίπεδο θα πρέπει πάντα να υπερισχύει του χαμηλότερου, εκτός ε, εάν υπάρχουν ε, ρήτρες εξαίρεσης στο υψηλότερο επίπεδο. Άλλα μέλη της ομάδας θεώρησαν ότι η αρχή της επικουρικότητας θα είναι σημαντική στον τομέα αυτών. Συμφωνίες που έχουν συνάψει ήδη οι εργαζόμενοι αναγκαστικά είναι πιο σημαντικοί και θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα σε σχέση με συμφωνίες σε υψηλότερο επίπεδο. Από την άλλη, καταλήξαμε σε συμφωνία όσον αφορά διάφορε παραμέτρους στι συλλογικέ συμβάσει. Για παράδειγμα, τη χρονική κάλαψη. Με το που λύγει μια τέτοια συμφωνία, τα μέλη της ομάδας θεώρησαν ότι οι παράμετροι θα πρέπει να καθορίζονται από τους ίδιους τους κοινωνικούς εταίρους κατά την συζήτηση της συλλογικής ε, σύμβασης. και σε περίπτωση που δεν καταλήξουν σε συμφωνία οι εταιροί, ο νόμος θα πρέπει να καθορίζει τις παραμέτρους που θα εφαρμοστούν. Για παράδειγμα, ε, παράταση εξαμηνιαία, κάλυψη όλων των προτύπων εργασίας στη συμφωνία, καθώς και τρίμηνη ε, προθεσμία για την απόρριψη της συμφωνίας. Τέλος, για να φτάσω στις δύο τελευταίες συστάσεις. Υπήρξε επίσης σε συμφωνία όσον αφορά το ρόλο της διαιτησίας. Τι μπορεί να γίνει σε περίπτωση που ε, τα μέρη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το περιεχόμενο συλλογικής σύμβασης τα μέλη της ομάδας θεώρησαν ότι θα πρέπει να εξετάζεται η διαιτησία, η διαμεσολάβηση, ως ε, ίστατη λύση, όχι όμως ως κοινή πρακτική. Ωστόσο, τα μέλη της ομάδας επίσης ε, επεσήμαναν ότι κάποιες προσαρμογές έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα, ε, εκ των οποίων κάποιες έχουν αναστραφεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας και ότι θα πρέπει να εξεταστούν αυτέ οι προσαρμογέ προτού υποβάλουμε συστάσει για συγκεκριμένε τροποποίησει. Η σύσταση μα υπαριθμών 11. Επίση, αποτέλεσε αντικείμενο συνένεση και αναφέρεται στη σημασία του κοινωνικού διαλόγου. και των συλλογικών διαπραγματεύσεων που μπορούν να αποτελέσουν πολύ σημαντικό μέσο για οικονομική ανάπτυξη και την προώθηση της απασχόλησης. Θελήσαμε να τονίσουμε τη σημασία της ενίσχυσης του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Και ε, φτάνω στην τελευταία σύσταση στην οποία θα αναφερθώ σήμερα. Ε, έχει να κάνει με το ρόλο της ε, δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης. Περίοδοι ανεργίας μπορεί να είναι αναπόφευκτες ακόμα και σε ε, υποανάπτυξη. Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, τα γραφεία έβρεση εργασίας, μπορούν να παράσχουν σημαντική αξία όσον αφορά την καλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. Ε, τα μέλη της ομάδας θεώρησαν ότι η περαιτέρω ενίσχυση της ε, δημόσιας αυτής υπηρεσίας για την κινητοποίηση των ανέργων αλλά και για την η εισαγωγή καλό, καλ, καλοσχεδιασμένων ε, ενισχύσεων ε, μπορεί να ε, βοηθήσουν την, το μέλλον της ελληνικής αγοράς εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Κύριε Μάρτινς, θα δώσω το λόγο τώρα εφόσον επιθυμείτε να θέσετε ερωτήσεις στον προσκεκριμένο μας, σε εσάς κυρία Γιονγκέριου. Ζητώ συγγνώμη, έχασα το πρώτο μέρος της ομιλία σας γιατί ήμουν απασχολημένη σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. Όμως, διαρωτώ με, εάν αν έχετε κάνει συγκεκριμένες συστάσεις για το καθεστώς των γνωμοδοτήσεων σας. διότι η επανεισαγωγή του κοινωνικού διαλόγου και οι στις συλλογικές συμβάσεις ε, βρίσκεται υψηλά στην ημερήσια διάταξη της σημερινής ελληνικής κυβέρνησης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από ό,τι ακούμε εμείς τουλάχιστον, λέει ότι δεν το θέλει αυτό, διότι αυτή υπήρξε μοναδική πραγματική μεταρρύθμιση στην ε, ελληνική οικονομία. Μπορούν όντως οι συστάσει να παραμεριστούν τόσο εύκολα και αυτά που ακούμε εδώ εμείς από τη δική μας Επιτροπή Απασχόλησης. Εγώ, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά θεμέλια της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην Ευρώπη. Πώς μπορούμε να πιέσουμε ώστε να γίνουν αποδεκτές οι συστάσεις σας. Έχετε κάποια στρατηγική προσέγγιση εσείς γι' αυτό. Αυτό θα μας βοηθούσε, εάν μπορούσατε να μας πείτε. Ε, τώρα η κυρία Τζιν Λάμπερτ για ερώτηση. Ευχαριστώ. Η δική μου ερώτηση είναι κάπως παρόμοια. Ποιες νομίζετε ότι θα είναι οι επιπτώσεις εάν εφαρμοστούν οι συστάσεις σας. Θεωρείτε ότι θα ενισχυθεί έτσι η αγορά εργασίας και θα αποκτήσει μια στέρεα βάση για τις μελλοντικέ εξελίξεις ή όχι. Όσον αφορά επίσης τις ικανότητες για παράδειγμα της, ε, των δημοσίων υπηρεσιών, επίσης διαιτησιών. Αυτά τα πράγματα ε, είναι τέλεια ή υπάρχει ανάγκη λήψος συγκεκριμένων μέτρων, μέτρων ώστε να γίνουν λειτουργικά τα πράγματα αυτά. Ή τέλος πάντων οι αλλαγές που θα επέλθουν να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Επίσης ε, ρωτώ εάν θεωρείται, εμείς έχουμε έχουμε κάνει μια συζήτηση, και κάναμε πριν δηλαδή, για την ε, βιομηχανία ενδύματος. Θεωρείτε ότι εκεί πρέπει να γίνει ακόμα κάποια δουλειά για να προωθηθεί. Ψάχνω να βρω κάποιους διπλωματικούς τρόπους για να εκφραστώ τώρα. Ε, πάντως έχει υποστεί ας πολύ σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Για να μην πω ότι έχει καταστραφεί. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας σχετικά με το τι είναι δυνατόν και τι όχι. Εμένα δεν μου φαίνονται τόσο κατάλληλες οι συστάσεις σας Και πάντως ε, διερωτώ με εάν σας έχουν στηρίξει ε, οι διάφοροι θεσμοί ή απλώς κάποιος σας έβαλε εκεί να λέτε αυτά που θέλει. Θα ακούσουμε και μια τρίτη ερώτηση από Φουντούλη. Έχει το λόγο κύριε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως είμαι και ο, ο μόνος Έλληνας εδώ Ευρωβουλευτής. παρότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό που συζητάμε εδώ. Μιλάμε για τις μεταρρυθμίσεις στην ελληνική αγορά εργασίας. Θα ήθελα να ρωτήσω ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις, όπως τις έχετε απαριθμίσει μία-μία εδώ, πιστεύετε ότι θα φέρουν στην Ελλάδα περισσότερες θέσεις εργασίας, θα φέρουν ανάπτυξη ή θα χειροτερεύσουν την κατάσταση. Συγκεκριμένα, μη είπατε στο, στην παράγραφο 4 για τη μερική απασχόληση ότι υπήρχε συνένεση για να μπορούν οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν τις κρίσεις. Σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται το δικαίωμά τους για μερική απασχόληση και ευέλικτες μορφές απασχόλησης και απολύουν τους εργαζομένους οι οποίοι είχαν πλήρες ωράριο και παίρνουν με τετράωρα εργαζόμενους και στην ουσία αυτοί οι άνθρωποι αντί για τέσσερις ώρες δουλεύουν έξι και οχτώ πολλές φορές. Και, με το πρόσχημα ότι αν δεν σας αρέσει φύγετε, θα έρθει κάποιος άλλος. Εν τω μεταξύ αυτή η ευέλικτη, μορφή απασχόληση κάνει και μεγάλη ζημιά στα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί οι ασφαλιστικέ φορές είναι πολύ λιγότερε, οι οποίε δίδονται στο, στο κράτος. Για το ελάχιστο ημερομίσθιο είπατε ότι δεν υπήρχε συμφωνία και κάποιοι έλεγαν ότι παίρνουν λιγότερα οι νέοι. Γιατί να παίρνουν λιγότερα οι νέοι. Για την ίδια προσφορά εργασία να αμείβονται διαφορετικά οι νέοι. Οι ανάγκε του είναι ίδιε, μην πω και περισσότερο. Και οι νέοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Κανεί δεν δουλεύει από χόμπι. Όλοι δουλεύουν για να επιβιώσουν και να περνούν και να ζουν αξιοπρεπώς. Οι συλλογικέ συμβάσει ε, και οι πρακτικές παράτασεις, δυστυχώ στην Ελλάδα οι συλλογικέ συμβάσει εργασία είναι πάρα πολλά χρόνια που έχουν καταργηθεί και δεν εφαρμόζονται και αυτό βεβαίω είναι ει βάρο των εργαζομένων γιατί δεν έχουν δικαιώματα να διεκδικήσουν. Όποιες μορφές απεργίας γίνονται είναι κατευθυνόμενες και δεν έχουν ουσιαστικά αποτέλεσμα γιατί γίνονται για να γίνονται, όχι για να κερδιθεί κάτι. Και με αυτή την κυβέρνηση που έχουμε στην Ελλάδα, φυσικά η οποία υποτίθεται ότι ήταν υπέρ της εργατικής τάξης, έχει κλείσει τα αυτιά της και δεν ακούει τα, αυτά που ζητάνε οι εργαζόμενοι. Ε, ο ΑΕΔ ναι, πιστεύω ότι μπορεί να παράσχει υπηρεσίε σαν αναβαθμιστεί. Πρόσφατα είχαμε πάει στη, με την Επιτροπή, δυστυχώ ήμασταν λίγοι ευρωβουλευτέ, στο, στο Κέλν και είδαμε εκεί μια δουλειά που γίνεται μεταξύ Γάλλων και Γερμανών και προσφέρονται θέσει εργασία ε, με μετακίνηση εργαζομένων από τη μία χώρα στην άλλη και έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει φαντάζομαι και στην Ελλάδα. Αυτά δεν θέλω να πω. Περιμένω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Ε, δεν είστε ο μόνος Έλληνε Ευρωβουλευτής, κύριε Φουντούλη. Υπάρχει και η κυρία Κούνεβα. Είναι εδώ κοντά μας και η κυρία Κούνεβα. Αν θέλετε κι εσείς τώρα λοιπόν να κάνετε την ερώτησή σας κυρία Κούνεβα, να δώσουμε μετά την ευκαιρία στον κύριο Μάρτιν να απαντήσει. Έχει το λόγο κύριε Κούνεβα. Αγαπητέ κύριε Μάρτινς, χαίρομαστε ιδιαίτερα που είστε σήμερα μεταξύ μα, ανάμεσα μας. Θα θέλαμε να, να μας λύσετε απορίε που έχουν να κάνουν με την διαδικασία αλλά και με την ουσία. Ω προ την διαδικασία, θα θέλαμε πραγματικά να γνωρίζουμε ποια είναι η προσθετέμενη αξία της πολύ σημαντικής δουλειάς που έχετε κάνει. Τι εννοώ με αυτό. Μια ομάδα σημαντικών επιστημόνων έχει εργαστεί για να εξετάσει ποιε είναι οι καλύτερες πρακτικές στην Ευρώπη σε σχέση με τα εργασιακά. Η αξιολόγηση που κληθήκατε να κάνετε αφορά την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο. Το μοντέλο που θα ακολουθήσει η Ευρώπη για την Ελλάδα είναι βεβαίο πως είναι το μοντέλο το οποίο θα επιβληθεί και σε άλλες χώρες. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε σε ποιο βαθμό τα συμπεράσματά σας θα ληφθούν υπόψη. Γνωρίζετε σε ποιο βαθμό θα υπερασπιστείτε τη δουλειά σας όταν μάλιστα ανήκετε με όλο σεβασμό στην εμπειρία σας, στην ομάδα της μειοψηφίας ως προς τις θέσεις που υιοθέτησαν. Ως προς την ουσία τώρα, αν και η διαδικασία στην οποία αναφέρθηκα πριν στηρίζει την ουσία Αναφέρομαι σε κάποια από τα συμπεράσματα της έκθεσής σας. Οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις αποτελούν πάγια πρακτική στα κράτη-μέλη. Αυτή η θέση στηρίζεται και από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και θα πρέπει να επανέλθει και στη χώρα μου εφόσον καλύπτεται από αυτές το 50% ενός κλάδου διάρκεια τους επίσης λέτε πως πρέπει να κατορίζεται από τους κοινωνικούς εταίρους. Στο θέμα της διατησίας επίσης αναλαμβάνει το κράτος μόνο όταν οι κοινωνικοί εταίροι δεν φτάνουν σε συμφωνία. Οι ατομικές συμβάσεις δεν μπορούν να προβλέπουν όρους χειρότερους από τις λογικές στις σωματικές απολύσεις έχει αποδειχτεί και από έρευνες στο ΩΣΑ ότι δεν τονώνουν την ανταγωνιστικότητα. Η Ελλάδα επιμένει στην προέγκριση της ομαδικής απολύσεις. Δεν έχει κρυθεί ακόμα το θέμα στο δικαστήριο. Ποια πιστεύετε πώς θα είναι η αποτελεσματικότητα μιας σκληρής εφαρμογής των ομαδικών απολύσεων. όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, μια από τις λύσεις που προτείνεται, αλλά που υπερασπίζεται όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, είναι να καθορίζουν οι το μισθό αυτό. Θα ήθελα να γνωρίζω αν έχετε και γιατί αντιρρήσεις επ' αυτού. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Άρα κύριε Μάρτινς έχετε τέσσερις ερωτήσεις ή μπορεί να πει κανείς ότι ήταν και πολιτικές τοποθετήσεις βέβαια από τις κυρίες Λάμπερ, τον κύριο, τον κύριο τον κύριο Φουντούρη, την κυρία Κούνεβα κλπ. Έχετε εσείς το λόγο τώρα και αν θέλετε, ε, μάλλον εγώ ε, ε, ε περιμένω μεγάλο ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας απηχούν και τις συζητήσεις που έχουν γίνει και στην ομάδα μας σε όλη αυτή τη δικασία των έξι μηνών. Αν, αν μου επιτρέπετε να ακολουθήσω την αντίστροφη σειρά και να αρχίσω με την τελευταία ερώτηση για τα αποτελέσματα, για τις απόψεις που έχουμε ακούσει από τους κοινωνικούς εταίρους στην Ελλάδα αλλά και αλλού η προστιθέμενη αξία της δικής μας δουλειάς μπορεί να είναι ωστόσο σημαντική με την έννοια ότι εμείς προσεγγίζουμε τα κρίσιμα αυτά θέματα από μια διεθνή σκόπια. Εργαστήκαμε πολύ σκληρά προβληματιζόμενοι στην βάση των εμπειριών μας από τις χώρες μας αλλά και στη βάση ενός μεγάλου αριθμού μελετών για να κάνουμε συστάσεις που να έχουν μεγαλύτερη χρησιμότητα και να επιτρέψουν η Ελλάδα να προχωρήσει. Ένα θέμα που αναγνωρίζω αμέσως είναι ποιες μπορούν να είναι οι βέλτιστες πρακτικές. Δηλαδή κάτι που μπορεί να είναι βέλτιστη πρακτική σε κάποιες χώρες μπορεί να μην είναι βέλτιστη πρακτική για άλλες χώρες. Υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που θα αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες χώρες και θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον σχεδιασμό των βέλτιστων ας πούμε θεσμών της αγοράς εργασίας στη συγκεκριμένη εκείνη περίπτωση. Θεωρούμε λοιπόν εμείς μέσα στις συστάσεις μας να λάβουμε υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζει επί του παρόντος η Ελλάδα. Επίσης προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι οι θεσμοί της αγοράς εργασίας μπορεί να υπόκειται και σημαντικές διαδράσεις, interactions δηλαδή, να υπάρχουν δηλαδή ομάδες χαρακτηριστικών σε ό,τι αφορά απολύσεις, σε ό,τι αφορά συλλογικές διαπραγματεύσεις, σε ό,τι αφορά ε, υπηρεσίες απασχόλησης. Πρέπει όλα αυτά να ε, ε, συζητούνται και να εξετάζονται ως σύνολο και όχι αναπερίπτωση. Αυτά χρειάζονται βέβαια βαθιά γνώση των ιδιαίτερων συνθήκων της κάθε χώρας στην περίπτωση της Ελλάδος θεωρήσαμε ότι η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του εργαζόμενου και οι συνθήκες για περισσότερη ευκαμψία μέσα στην οικονομία, ίσως εκεί υπήρχε κάποιος χώρος βελτίωσης και εντοπίσαμε ένα συγκεκριμένο τομέα στον οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως και που είναι ο χώρος των ομαδικών απολύσεων και που θεωρήσαμε ότι υπήρχε μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις πρακτικές που ισχύουν στην Ελλάδα και στις πρακτικές που ε, διαπιστώνονται σε, στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία των άλλων χωρών μελών. Εκεί θεωρήσαμε λοιπόν ότι για να προχωρήσει μπορούσαν να γίνουν κάποιες προσαρμογές, δηλαδή να μειωθεί η απέτηση διοικητικών πράξεων για να επιτραπούν οι ομαδικές απολύσεις. Θεωρήσαμε ότι εκεί υπήρχε χώρος αλλαγής. Από την οικονομική σκοπιά εμείς θεωρήσαμε ότι οι περιορισμοί στις ομαδικές απολύσεις μπορεί εν τέλει να παίξουν τον ρόλο των του περιορισμού των επενδύσεων που θα κάνουν κάποιες επιχειρήσεις. Και η ελληνική οικονομία αναμένει, καίγεται για επενδύσεις από επενδυτικές πηγές και κυρίως από διεθνείς επενδυτικές πηγές. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τους όρους αυτούς, κάτι τέτοιο, μια τέτοια αλλαγή μπορεί να ε, δείξει ότι η χώρα επιθυμεί να προσελκύσει ε, σημαντικές επενδύσεις. Βέβαια, τούτου λεχθέντος η ομάδα μας και τα μέλη της είπαν σαφώς ότι αναγνωρίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, ότι οι προκλήσεις αυτές είναι πολύ περίπλοκες και ότι με πολλούς τρόπους έχουν και πολλές πτυχές. Υπάρχουν πολλά θέματα που προέρχονται από την αγορά προϊόντων, από διάφορα γεγονότα τα οποία συνέβηκαν τα τελευταία χρόνια και που μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντικά για να εξηγηθούν οι τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και η αγορά εργασίας της Πάντως, εμείς θεωρούμε ότι η υιοθέτηση ορισμένων συστάσεών μας, αλλά και μια περαιτέρω συζήτηση για ιδιαίτερου τομεί που δεν σημειώθηκε συνένεση, μπορεί να βοηθήσει ωστόσο για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία και στην αγορά εργασίας της. Έρχομαι τώρα στην τρίτη με τη σειρά ερώτηση του κύριου Φουντούλη δηλαδή, Πράγματι, θίξατε σημαντικά θέματα. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσω να, ε, να απαντήσω σε όλα. Μία συγκεκριμένη ερώτηση που κάνατε είναι σε ποιο βαθμό είναι κατάλληλο, είναι σωστό δηλαδή, οι νεαροί εργαζόμενοι να λαμβάνουν χαμηλότερο μισθό. Βεβαίω, εμεί θεωρούμε ότι οποιοδήποτε και ανεξαρτήτω ηλικία ή ανεξαρτήτω άλλων χαρακτηριστικών θα πρέπει να ε, γίνεται αντικείμενο ισότιμης μεταχείρισης. Ένα θέμα ωστόσο για τον κατώτατο μισθό είναι ότι μπορεί να υπάρχει ένας ισχυρός συσχετισμός ανάμεσα στην ηλικία και στην εμπειρία στην αγορά εργασία. Και με τον τρόπο αυτό εννοούμε και την παραγωγικότητα. Εάν δηλαδή ο εργοδότης λαμβάνει μια απόφαση σχετικά με την επιλογή που θα κάνει ποια παραγωγικότητα μπορεί να αναμένει από τον εργαζόμενο και τι μισθό θα του πληρώσει, εάν βάλει κανείς τον ίδιο κατώτατο μισθό για όλους τους εργαζόμενους, μπορεί αυτό τελικά να οδηγήσει σε αρνητική μεταχείριση ορισμένων νεαρών εργαζόμενων, αφού θα θεωρήσει ο εργοδότης ότι οι νεαροί αυτοί εργαζόμενοι δεν έχουν τις ίδιες δεξιότητες, δεν έχουν την ίδια επαγγελματική εμπειρία και δεν μπορεί να λάβει τα ίδια βάρη αν βάλει κανείς έναν κατώτατο μισθό που θα είναι υπερβολικά υψηλός συγκρινόμενος με την παραγωγικότητα του εργαζόμενου, τότε θα έχει αρνητικές επιπτώσεις. Και θα αποβιώθω σε βάρος πολλών εργαζόμενων νεαρής ηλικία. Γνωρίζουμε δε ότι η ανεργία των νέων στην, ε, ε, στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλή και φτάνει και το 40%. Αυτά σκεφτόντουσαν ορισμένα μέλη της ομάδας μας άλλα μέλη της ομάδας μας θεώρησαν ότι είναι προτιμητέα μια άλλη προσέγγιση. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την μείωση του κατώτατου του μισθού, σε ό,τι αφορά την συντόμευση των περιόδων που θα καταβάλλεται ο χαμηλότερος μισθός στις ομάδες αυτές εργαζόμενων και ούτω καθεξής. Με ρωτήσατε και για τις συλλογικές συμβάσεις και σε ποιο βαθμό επιβάλλονται τι ρόλο παίζουν στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου. Αυτό ήταν πράγματι ένα θέμα το οποίο αντιμετώπισαν διαφορετικά τα διάφορα μέλη της ομάδας. Πάντως όλα τα μέλη της ομάδας εξετίμησαν την ε, δυνητική σημασία των συλλογικών συμβάσεων. Ένα θέμα το οποίο ανησύχησε ορισμένα μέλη της ομάδας ήταν θέματα αντιπροσωπευτικότητας ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού εργατικού δυναμικού δεν είναι μέλη ε, εργατικών συνδικάτων. Πολλά μέλη, ε, πολλοί εργαζόμενοι δηλαδή επιχειρήσεων δεν είναι μέλη συνδικάτων. Αυτό εξηγείται από ορισμένου παράγοντες, για παράδειγμα και από το μικρό μέγεθος των περισσότερων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αυτό αποτελεί όντως πρόκληση. Σε ποιο βαθμό δηλαδή μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις που ωστόσο δεν βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό αντιπροσωπευτικότητας μπορεί ενδεχομένως να αποτελέσουν πρόβλημα για την πλήρη προσαρμοστικότητα της ελληνικής αγοράς εργασίας. Βέβαια, η Ελλάδα έχει σημαντική εμπειρία συλλέξει τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου αντιπροσωπευτικότητας, δηλαδή αντιπροσώπευσης των εργαζόμενων με ενώσεις προσώπων που αποδείχθηκε τελικά πολύ επιτυχημένο μοντέλο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη παρά τις αυστηρού τους αυστηρούς περιορισμούς αντιπροσωπευτικότητας, για παράδειγμα για μια ένωση προσώπων, για να μπορέσει να κάνει μια συλλογική σύμβαση με τον, με τον εργοδότη, λέει ότι θα πρέπει τουλάχιστον τα τρία πέμπτα να είναι μέλη. Αυτό είναι ένα νέο μοντέλο το οποίο έχουν επικρίνει ορισμένοι ενδιαφερόμενοι και ιδίω τα συνδικάτα, αλλά ίσως έπαιξαν ένα ρόλο ε, στο να δημιουργηθεί ένας μεγαλύτερος δυναμισμός για τις ε, συλλογικές συμβάσεις, υπέρ των συλλογικών συμβάσεων, αν και ίσως με κάποιο διαφορετικό τρόπο από ό,τι ε, συνέβαινε στην Ελλάδα μέχρι το 2011. Για την προηγούμενη τώρα από τη δική σας ερώτηση, Δυστυχώς δεν έχω σημειώσει το όνομα της ε, Ευρωβουλευτού. Α, η κυρία Λάμπερτ. Η κυρία Λάμπερτ, λοιπόν, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της ενδεχόμενης εφαρμογής των συστάσεών μας. Εμείς ε, έχουμε την πεποίθηση ότι οι συστάσεις αυτές μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην βελτίωση ορισμένων δικτών της αγοράς εργασίας, παρόλο που αντιλαμβανόμαστε ότι τα προβλήματα είναι πολύ πιο περίπλοκα και βεβαίως ότι η αγορά εργασίας είναι μία συνιστόσα μόνο από τις πολλές της ελληνικής οικονομίας. Αναφερθήκατε ειδικά στον ρόλο των δημοσίων υπηρεσιών ως εργοδότου και στην διαιτησία. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ την υπηρεσία δημόσιας απασχόλησης και ορισμένα κέντρα στην χώρα και ευχαριστώ ιδιαίτερα την ελληνική κυβέρνηση που με επέτρεψε να επισκεφθώ τα μέρη αυτά. Είδα τις σημαντικές βελτιώσεις που εφαρμόζονται πράγματι εκεί. Νομίζω ότι πρόκειται για σημαντική πρόοδο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Οι υπηρεσίε αυτές έχουν γίνει όλο και πιο ισχυρές σε ό,τι αφορά την ε, δυνατότητά τους να ενισχύσουν τους ανέργους Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν, ε, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη να προωθηθεί περισσότερο και όπως λέμε και στην εκθεσή μας, θεωρούμε ότι χρειάζονται και άλλες προσπάθειες ό,τι αφορά την παρακολούθηση της εξέλιξης των ανέργων, ε, να προωθηθούν και ε, νέες πολιτικές απασχόλησης. Υπάρχουν και ορισμένες πρόσφατες συστάσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η προσφορά ε, περισσότερη στήριξη σε αυτούς που είναι μακρόχρονα άνεργοι. Ε, έχει γίνει λοιπόν κάποια πρόοδο, και σε ό,τι αφορά τι ε, βέλτιστες πρακτικέ, αλλά και πολλέ χώρες μέλη έχουν ενισχύσει πολύ σημαντικά, έχουν επενδύσει πολύ σημαντικά τι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης με αποτελέσματα. Έχουμε το παράδειγμα του Ενωμένου Βασιλείου από τη μια, της Γερμανίας από την άλλη, που είναι περιπτώσεις που νομίζω ότι δείχνουν κάποιον ενδιαφέρον, δίνουν κάποιον ενδιαφέρον για την σκοπιά αυτή των βέλτιστων πρακτικών. Φτάνω τέλος στην πρώτη σας ερώτηση. που στράφηκε γύρω από το δυναμικό των συστάσεων μας, τον ρόλο του κοινωνικού διαλόγου και της επανεισαγωγής του στην Ελλάδα, γιατί είναι διάσταση στρατηγικής που προκύπτει από τις συστάσεις που έχουμε κάνει. Νομίζω ότι κατανοώ την ερώτησή σας και τη βρίσκω ενδιαφέρουσα και σημαντική. Η δική μας οι δικές μας απόψεις ως εμπειρογνωμόνων προέρχονται από τις εμπειρίες που έχουμε συλλέξει, από τις συζητήσεις μας και έχουμε κάνει ορισμένε συστάσεις. Η άποψή μας ήταν περισσότερο αυτή του πανεπιστημιακού, που δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενος στην ε, διαμόρφωση πολιτικής. Υπάρχει, υπάρχει απόσταση μεταξύ των δύο χώρων, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν προσεγγίσει πάρα πολύ οι δύο αυτοί κόσμοι. Και νομίζω ότι αυτό βέβαια είναι προς όφελος όλων αλλά κατανοώ ότι ορισμένες από τις ε, συστάσεις αυτές έγιναν ευμενώς δεκτές από τους κοινωνικούς εταίρους, θέματα για παράδειγμα για την επανεισαγωγή μηχανισμών επέκτασης, αυστηρά κριτήρια αντιπροσώπευσης, αυτά έγιναν όπως είπα ευμενώς δεκτά, οι πρακτικές επέκτασης υποστηρίχθηκαν και στην Ελλάδα από το 2012, και ήταν μια σημαντική αλλαγή. Οι κοινωνικοί εταίροι ίσως θα ήθελαν να έχουν και περισσότερο λόγο σε ό,τι αφορά τον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Όπως είπα, η ομάδα μας ήταν διασπασμένη στο θέμα αυτό. Ορισμένοι από τα μέλη μας θεώρησαν ότι αυτό πρέπει να είναι ευθύνη της κυβέρνησης. ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει και τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις ενό κατώτατου μισθού που θα ε, θεσπιζόταν σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Η δυσκολία είναι πάντοτε να βρεθεί ποιο είναι το καλύτερο επίπεδο του κατώτατου μισθού, ώστε ο κατώτατο μισθό εφόσον αυξηθεί σε ένα ποσοστό που είναι υπερβολικά υψηλό, θα έχει αυτομάτως αρνητικέ επιπτώσεις στην απασχόληση. Η πρόκληση λοιπόν είναι να βρεθεί η σωστή ισορροπία στην θέσπιση του κατώτατου μισθού, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η ενδεχόμενη θετική επίπτωση στην αγορά εργασία χωρί να μεγιστοποιηθεί η ενδεχόμενη αρνητική επίπτωση στην αγορά εργασία. Προσπαθώντας να συνοψίσω θα έλεγα ότι οι συστάσεις αυτές μπορούν να είναι σημαντικές και όχι μόνο για την Ελλάδα. Μπορούν να βοηθήσουν να γίνει και άλλη συζήτηση και σε ό,τι αφορά ενδεχόμενε προσαρμογές σε θεσμούς των αγορών εργασίας και σε άλλες χώρες αφού βασίζονται σε εμπειρίες από την πράξη και σε μια σύγκριση των θεσμών μας σε μια συγκεκριμένη χώρα μέλος με αυτές των άλλων χωρών, προσπαθώντας να ε, θεσπίσουμε τις ε, καλύτερες πρακτικές. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να έχει σημαντικό ενημερωτικό χαρακτήρα και να διαμορφώσει πολιτικές. Διότι εγώ θεώρησα ότι ήταν μεγάλη ευκαιρία για τα μέλη της ομάδας μας και ε, και ήμασταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που μπορέσαμε να συμβάλλουμε στην διαδικασία αυτή και να προσφέρουμε συστάσεις και στην ελληνική κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μπορέσουν να τις ενσωματώσουν, να ενσωματώσουν στις πρακτικές που θα θεωρήσουν κατάλληλες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η κυρία Κούνεβα είχε μια επιπρόσθετη ερώτηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μπερδευτεί. Από τη μία λέτε πως κάτι που μπορεί να είναι καλό για μια χώρα δεν σημαίνει πως είναι και για μια άλλη. Απ' την άλλη λέτε πως οι σημαντικές απολύσεις στην Ελλάδα γίνονται με πολύ διαφορετικό τρόπο από τις άλλες χώρες και αυτό το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Όπως σας είπα, μελέτες του ΟΑΣΑ για την Ελλάδα αποδεικνύουν πως οι ομαδικές απολύσεις δεν συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Πού στηρίζετε λοιπόν αυτά που μας λέτε. Και η κυρία Γιονγκέριους, έχει, έχει μια ερώτηση. Ναι, μια ερώτηση υπομορφή συνέχειας. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων ενημερώθηκε μετά από επικρίσεις από διάφορες ε, πλευρές σε σχέση με τη δράση της Τρόικας στην Ελλάδα η οποία ασχολήθηκε μόνο με το δημοσιονομικό σκέλος του μνημονίου και με τίποτα άλλο. Και όταν αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων χρειάστηκε να μιλήσει για τις βέλτιστες πρακτικές για κοινωνικά ζητήματα, για την ελληνική κυβέρνηση, αυτό ε, ίσως θα σήμαινε ε, ότι ζητάτε μια συγνώμη για, για το πολύ επαχθές πρόγραμμα που επιβλήθηκε στην Ελλάδα. Τώρα εσείς μας λέτε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι εκείνη που θα δει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Δεν εξαρτάται όμως και από την Τρόικα η οποία θα πρέπει να δώσει μια απάντηση, να ανταποκριθεί στην έκθεσή σας ή έστω να αποκριθεί. γιατί η ελληνική κυβέρνηση ίσως ε, τάσεται υπέρ των προτάσεών σας, αλλά είναι μια χώρα υπό πρόγραμμα. Και γι' αυτό υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παρισφρίουν και η Τζιν και εγώ επισκεφτήκαμε το Μπαγκλαντές τρεις εβδομάδες πριν και λέγαμε ακριβώς κάναμε κήρυγμα ότι δεν έχουν ε, εργατικό νόμο που να συμβαδίζει με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και τις ε, συναφείς συμβάσεις. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση που, μια χώρα μάλλον, που ανήκει και στην Ευρωζώνη. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με τη δική σας πρόταση. Δηλαδή δεν αρκεί να πείτε ότι επαφιέμεθα στην ελληνική κυβέρνηση για να κάνει κάτι. Ευχαριστώ, Άγνες. Ο κύριος Σαβιανόπουλος έχει το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μαρτένση, μιλάτε ε, σαν μέρος της Επιτροπής των ε, Εμπειρογνωμόνων, η οποία υποτίθεται ότι στηρίχθηκε πάνω σε αυτό που ονομάζεται βέλτιστες πρακτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις πρακτικές του ILO. Το πιστεύω αυτό, έτσι είναι τα πράγματα. Απλώς θέλω να ξέρω αν έχει συνέστηση η Επιτροπή για τα εξή που θα σας πω παρακάτω. Πρώτον ότι η μείωση του μέσου μισθού στην Ελλάδα, του μέσου μισθού, όχι των κατώτερων, όλα τα τελευταία χρόνια είναι πάνω από 40%. Δεύτερον, ότι οι απολύσεις ε, έχουν φτάσει το επίπεδο της ανεργίας στο 1,5 εκατομμύριο ανέργων. Και επίσης να προσθέσω από τους υπόλοιπους εργαζόμενους τυπικά εργαζόμενους, το 1 εκατομμύριο είναι απλήρωτοι από 8 έως 12 μήνες. Απλήρωτοι. Εργάζονται μένουν, δεν πληρώνονται δε. Στην πραγματικότητα έχουν την τύχη των ανέργων. Στην, ε, ε στο πόρισμα της Επιτροπής Απειρογρομώνων και ειδικά όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασία, Υπάρχουν τόσε εξαιρέσει μέσα, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση μια επιχείρηση, ότι μπορεί να κατεβάσει τον μισθό ε, ανάλογα με τι δυσκολίε τη που τελικά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σύστημα συλλογικών συμβάσεων εργασία παρά μόνο η διαπίστωση ότι μια εταιρεία μπορεί να έχει κάποιε οικονομικέ δυσκολίε και να κατεβάζει από μόνη του μισθού. Τρίτον, ε, θεσπίζεται, σύμφωνα με το πόρισμα τη ε, Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, θεσπίζεται ο λεγόμενο υποκατώτατο μισθό, που σημαίνει ότι θα υπάρχουν μισθοί, που βεβαίω θα είναι πάρα πολλοί, οι οποίοι θα είναι κάτω από τον κατώτατο μισθό. Κάτι που υπήρχε μέχρι τώρα στην Ελλάδα, με βάση το μνημόνιο, δηλαδή οι νέοι κάτω από 25 χρονών, τώρα όμω αλλάζει η κατάταξη και λέει όσοι δεν έχουν εργασιακή εμπειρία. Αυτό σημαίνει, που και για του νέου ήταν καταδικαστέο και άδικο, σημαίνει ότι μπορεί να είσαι 30, 35, 40, 45 χρονών, να μην έχει εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο στο οποίο καλείσαι να δουλέψει και τελικά να αμυφθεί σε αυτή την ηλικία και με πολλά χρόνια εργασία πίσω, να αμυφθεί με τον υποκατώτατο μισθό, δηλαδή γύρω στα 250 με 300 ευρώ. Τέλος, ε, προφανώς γνωρίζετε ότι πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση έχει ε, θεσμοθετήσει και έχει απελευθερώσει πλήρως το καθεστώς των λεγόμενων φιλεμπορικών γραφείων. Δηλαδή γραφεία τα οποία ενοικιάζουν για χαμηλότατους μισθούς εργαζόμενους σε εργοδότες και ξέρετε εδώ υπάρχουν συγκεκριμένοι κλάδοι οι οποίοι ε, πώς το πω, έχουν ε, ξεπεράσει κάθε όριο. Συγκεκριμένα η κλάδη των εφοπλιστών ή των αυπηγοεπισκευαστών έτσι, που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τέτοια δουλεμπορικά γραφεία χρησιμοποιούν πολιτικό κόμμα που τα στείνει τη Χρυσή Αυγή οι οποίοι ξέρετε ότι για την ίδια υπόθεση έχει κάνει δολοφονικέ επιθέσει στην Ελλάδα και δικάζονται. Αυτό, αυτό είναι με κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίω με συμφωνία και τη ελληνική κυβέρνηση, τα δουλεμπορικά γραφεία. Το ξέρετε αυτό. Και τελευταίο, με τι ομαδικέ απολύσει. Ξέρετε ότι η Ελλάδα και άλλε χώρε, αλλά ειδικά η Ελλάδα, βρίσκεται σε μια αναδιάταξη των κλάδων. Άλλοι κλάδοι εξαφανίζονται, θέλουν άλλοι να ενισχυθούν. Ε, θα έχουμε μια μεγάλη αναδιάταξη. Αυτό σημαίνει ότι πολλέ επιχειρήσει θα κλείσουν. Άρα λοιπόν το ζήτημα των ομαδικών απολύσεων είναι, θα διευκολύνει κατά πολύ ε, δεκάδε χιλιάδε απολύσει, ούτω ώστε με πολύ μικρότερου μισθού, κυριολεκτικά ψίχουλα, να προσληφθούν για ελάχιστο χρονικό διάστημα κάποιοι άλλοι σε έναν άλλον κλάδο. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό θα πέσει το επίπεδο μισθών στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο και από το 40%. Συνοπολογισμένο και το εγγυημένο εισοδήματο, το βεβαίω είναι κυριολεκτικά ψίχουλα, 250 με 300 ευρώ. Τι λέτε για όλα αυτά, γιατί όλα αυτά συντείνουν και σα πιστεύω ότι είναι οι ευέλικτε πρακτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώ, συντείνουν σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση των μισθών στην Ελλάδα. Σα ευχαριστώ. I put Mr. Fontoulis on the list, but we'll start with... Θα αρχίσουμε με τις απαντήσεις. Ο κύριος Φουντούλης είναι επίση στον κατάλογο. Thank you very much. Um, Μετά θα πάρει το λόγο ο κύριος Φουντούλης. Ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο ερώτημα αφορά τις ε, μαζικές απολύσεις και τις σχέσεις με την απασχόληση. Γνωρίζω ότι διενεργήθηκαν πολλές μελέτες και από τον ΩΣΑ που ασχολούνται με αυτό το συσχετισμό Από όσο κατανοώ από τις μελέτες αυτές, εάν δούμε το ζήτημα με όρους ανεργίας, η μεγαλύτερη ευελιξία στις απολύσεις δεν συσχετίζεται άμεσα με τον δίκτυο ανεργίας. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ευελιξία και αν δεν υπάρχουν τα ίδια όρια και ο ίδιος συσχετισμός με τις ε, απολύσεις μπορεί να οδηγήσει και σε αύξηση των προσλήψεων αυτή η ευελιξία ενώ. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δούμε την δυναμική της ε, απασχόλησης υπάρχουν ε, φυσικά επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν, απολύουν, ψάχνουν νέους αγοραστές, έχουν νέους προμηθευτές και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει μία ε, μεταβλητή δυναμική. Και ως προς τις απολύσεις, συλλογικές σημεί και το δίκτυο ανεργίας έχουμε ενδεχομένως και τις περισσότερες προσλήψεις, διότι οι επιχειρήσεις μπορούν να προσλάβουν και περισσότερους εργαζόμενους πολλές φορές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν απολύσεις. Φυσικά και υπάρχουν. Αν δούμε όμως αυτό το συσχετισμό μεταξύ απολύσεων και μακροχρόνιας ανεργίας και όχι βραχυχρόνιας ή μεσοπρόθεσμης και των ευρημάτων ακόμα και του ΩΣΑ, βλέπουμε ότι υπάρχουν θετικές επιπτώσεις στην απασχολησιμότητα και την απασχόληση σε σχέση με τη μακροχρόνια απασχόληση. Γιατί εάν δεν υπάρχει περιοριστικό πλαίσιο έχουμε χαμηλότερα επίπεδα μακροχρόνιας απασχόλησης Δηλαδή είναι ευκολότερο να βρει κανεί εργασία αν και φυσικά υπάρχει υψηλό ποσοστό απολύσεων. Ίσως υπάρχει όμως μία αντιστάθμιση ενδεχομένως. Γίνεται όμως μία συζήτηση επί του θέματος για να δούμε εάν υπάρχουν και θετικές πτυχές ε, σε σχέση με τους κανόνες προσλήψεων για να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία για τη δημιουργία απασχόλησης. Αυτό αφορά και κίνητρα που δίδονται προς τις επιχειρήσεις για την πρόσληψη νέων εργαζομένων. Το δεύτερο ερώτημα αφορούσε την στρατηγική και τη σχέση μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και Τρόικας. Δηλαδή κατά πόσο αυτή η στρατηγική θα οδηγήσει σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Το θέμα αυτό είναι άκρος ενδιαφέρον, αλλά θέλω να κατανοήσετε ότι εδώ είμαι εμπειρογνώμονας από αυτή την Επιτροπή που χρειάστηκε να κάνει συγκεκριμένες συστάσεις ε, προς την αγορά εργασίας. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, γιατί οι απόψεις θα ήταν δικές μου και όχι της ομάδας την οποία εκπροσωπώ. Προτιμώ λοιπόν να απόσχω από την απάντηση αυτή της συγκεκριμένη ερώτησης, αν και κατανοώ ότι είναι άκρος σημαντική σε σχέση με τις μελλοντικές επιπτώσεις των συστάσεών μας. Η τελευταία ερώτηση αφορά τις τρέχουσες προκλήσεις της ελληνικής αγοράς και της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Έχω απόλυτη επίγνωση τη... για τις μεγάλες ανησυχίες που υπάρχουν από τον υψηλό δίκτυ ανεργίας. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που είναι και εκτός αγοράς εργασίας. Θα επανέλθω όμως σε κάτι που είπα πριν. Υπάρχει δυνατότητα βελτιστοποίησης των ε, πρακτικών και των βέλτιστων πρακτικών από πλευράς λειτουργίας της αγοράς και εκεί έχουμε κάνει συστάσεις. Αν και αυτό δεν απαντά σε πληρότητα στις ανησυχίες και τις προκλήσεις, υπάρχει μία στοχοθέτηση των μεταρρυθμίσεων και προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να συνεισφέρουν για να έχουμε χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας και υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης. Είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα και υπάρχουν πολλές προκλήσεις που ανακύπτουν από το παρελθόν. Αλλά νομίζω ότι πολλές από αυτές τις ε, μεταρρυθμίσεις θα διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο. Τώρα, ως προς τον χρονισμό των ε, μεταρρυθμίσεων. Ίσως θα υπήρχε καλύτερη εφαρμογή σε περίοδο ανάπτυξης και όχι σε περίοδο κρίσης, όμως τη στιγμή που δεν έγιναν πριν έχει μεγάλη σημασία η περίοδος προσαρμογής με την εφαρμογή αυτών των ε, μεταρρυθμίσεων. Καλύτερα νωρίτερα παρά αργότερα. Ο κύριος Φουντούλης έχει το λόγο. Ε, δεν μου απαντήσατε στην προηγούμενη ερώτηση που σας είχα κάνει για τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και τις οποίες εκμεταλλεύονται οι εργοδότες και απασχολούν τους εργαζόμενους. Υποτίθεται για τετράωρη απασχόληση και πολλές φορές τους απασχολούν ολόκληρο το ωράριο, το, το οχτάωρο δηλαδή, ε, ενώ πληρώνουν μισέ ασφαλιστικέ εισφορές με αποτέλεσμα να καταραίουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Όσο για τον εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού κόμματο, απαξιώνω το απαντήσω γιατί το εργοστάσιο έχει κλείσει και έχει μείνει ένα υποκατάστημα στην Ελλάδα που θα κλείσει και αυτό. Ευχαριστώ. Well, that was not... Δεν νομίζω ότι ήταν ερώτηση αυτή. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μας επισκεφτήκατε. Είμαι βέβαιη ότι θα επανέλθουμε και σε εσά και σε άλλους που προσπάθησαν να συμπαρασταθούν στην Ελλάδα και να βρουν λύσεις. Είναι πολλά τα μέλη της δικής μας Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό και γνωρίζω ότι Υπάρχουν δραστηριότητες σε πολλές πολιτικές ομάδες, όπως στη δική μου, την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Υπάρχει ενδιαφέρον για υποβολή νέων προτάσεων σε συνεχή βάση για να βρεθούν τρόποι να βρεθούν νέοι τρόποι για την Ελλάδα για παράδειγμα, να είναι δυνατόν να έχει ένα ισχυρό σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως είπατε επανειλημμένα κατά την εισαγωγή σας. Να βρεθούν τρόποι που να μην δίνουν την εντύπωση ότι θα χρειαστούν δεκαετίες ε, μέχρι να επανέλθει η Ελλάδα σε αξιοπρεπή τρόπο ζωής. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία, σας, για την παρουσία σας. Και είμαι αρκετά βέβαιη ότι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξή μας ε, και ελπίζω να μπορέσουμε να σας ξαναπροσκαλέσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Αυτό σημαίνει επίση ότι ολοκληρώθηκε η σημερινή μα συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρία θα πραγματοποιηθεί 8 Δεκεμβρίου ε, και θα είναι ολοήμερη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ για την ε, σημερινή παρουσία σας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.